είναι απαραίτητο να δούμε την συνολική ε, μεθοδολογία για τα ε, περιθώρια ασφαλείας και γενικά για όλο τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να μειώσουμε τους κινδύνους. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι μία χρονική περίοδος δύο ε, ημερών συσσωρεύει περισσότερο από θέμα ασφαλείας για τον κεντρικό αντισυμβαλόμενο από ότι σε μια μέρα. Αυτό σημαίνει ότι είναι κατά μία τετραγωνική ρίζα του 2, 41% δηλαδή, περισσότερο το ποσό που συσσωρεύεται σε δύο μέρες από ότι σε μία. Εμείς όμως έχουμε την μεθοδολογία αυτή που αναφέρεται ως χονδρική ε, ακαθάριστη συσσόρευση και κατάθεση του ποσού ασφαλείας για κάθε, ε, για κάθε, για κάθε συμβαλόμενο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει και το συμψηφισμό. Δηλαδή αν η έκθεση ενός ε, πελάτη του αντισυμβαλόμενου, κεντρικού αντισυμβαλόμενου ε, εξισώνει την ε, έκθεση κάποιου άλλου, τότε μπορεί να υπάρχει η κατάθεση ενός ποσού που είναι το συμψηφισμένο περιθώριο. Εμείς συζητούσαμε λοιπόν για την, ε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν το ποσό χωρίς συμψηφισμό για μια μέρα ήταν υψηλότερο από το ποσό δύο ημερών με συμψηφισμό. Αυτό ήταν και το αντικείμενο των συζητήσεών μα με τον Λόρδο Χίλ το Φεβρουάριο. Βάσει τη δική μα ανάλυση που χρησιμοποίησε πραγματικά στοιχεία 7 ημερών, προσπαθήσαμε να δούμε ποιο θα ήταν το απόθεμα ασφαλεία που θα απαιτεί για το καθεστώ το ευρωπαϊκό ή το αμερικανικό για τα 9 μεγαλύτερα μέλη τη Ένωση των Κεντρικών Αντισυμβαλωμένων στι ΗΠΑ που καλύπτουν 80% του συνολικού ποσού ασφάλεια. Αυτό που είδαμε είναι ότι το ποσό χωρίς συμψηφισμό για μία μέρα ήταν πολύ μεγαλύτερο από το ποσό δύο ημερών με συμψηφισμό για κάθε αποθετήριο και για κάθε μέρα. Επομένως, το συνολικό ποσό περιθωρίου που απαιτείται για μία μέρα χωρίς συμψηφισμό έφτανε το 421 ως μάξιμου του ποσού για δύο μέρες με συμψηφισμό και δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερο, μικρότερο από το 160% αυτού του ποσού. Και είδαμε και άλλες μεγαλύτερες διαφορές για άλλα ε, κεντρικά αποθετήρια. Συγγνώμη που σας τα παρουσιάζω αυτά που είναι τεχνικά, αλλά αυτό το οποίο θέλω να δείξω είναι ποιο είναι το αποτέλεσμα της χρήσης συμψηφισμού και της επιμήκυνσης του χρόνου ε, εκτέλεσης των εντολών αυτών. Έχω δύο διαγράμματα που δεν έχουν στοιχεία γιατί πρέπει να προστατεύσουμε την ε, εμπιστευτικότητα αλλά καταδεικνύουν καλύτερα τα θέματα αυτά. Ο πρώτος, το πρώτο γράφημα το οποίο βλέπετε δείχνει το αποτέλεσμα του συμψηφισμού συγκρίνοντας την ε, μία μέρα με συμψηφισμό με τη μία μέρα χωρίς συμψηφισμό. Εμείς φυσικά χρησιμοποιούμε δύο μέρες με συμψηφισμό, μία μέρα, ε, μία μέρα χωρίς συμψηφισμό, αλλά πήραμε χαρτοφυλάκια για τρία μέλη του, της Ένωσης των Αποθετηρίων και τα βλέπετε αυτά στον κατάλογο. Μπορείτε να δείτε ποιες είναι οι δυνατότητες να υπάρχουν συμψηφισμοί και θεωρούμε ότι για κάθε πελάτη το ποσό του ε, περιθωρίου ασφαλείας πρέπει να είναι, γύρω, 100 ευρώ και βλέπουμε ότι σε, την, αυτό το σενάριο παίρνει το κεντρικό αποθετήριο 3.000 δολάρια. Ενώ στη συνέχεια με το ίδιο, με τις ίδιες αρχικές ε, υποθέσεις, εάν επιτραπεί ο συμψηφισμός, θα πάρει το κεντρικό αποθετήριο μόνο 800 δολάρια. Βέβαια, όλα αυτά θα εξαρτώνται στην πραγματική ζωή από την σύνθεση των χαρτοφυλακίων. Και στο δεύτερο γράφημα χρησιμοποιούμε δύο ημέρες για τον συμψηφισμό έναντι μίας μέρας για τον ε, χωρίς συμψηφισμό. Και βλέπετε ότι στη δεύτερη περίπτωση με συμψηφισμό σε διάρκεια δύο ημερών φτάνουμε στα 1120 δολάρια. Δηλαδή υπάρχει η αύξηση 41% ρίζα 2 δια 1 δηλαδή, αλλά αυτό δεν αρκεί για να δισταθμίσει το αποτέλεσμα του συμψηφισμού. Έχουμε 3.000 έναντι 1.120 δολαρίων με τον συμψηφισμό. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια ακραία κατανομή των ε, θέσεων που κατέχουν οι συμβαλόμενοι για να μπορέσουμε να φτάσουμε τα 3.000. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν και την, τις ε, θέσεις οι οποίες μπορεί να είναι ανισομερείς. Επομένως, τι σημαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Λόγω εμπιστευτικότητας δεν μπορούμε να σας δώσουμε τα συγκεκριμένα στοιχεία για όλους τους ε, αντισυμβαλόμενους. Φυσικά αυτό το έχουμε συζητήσει με την Κομισιόν. Το τρίτο, ο τρίτος, ε, τρίτο γράφημα δείχνει το αρχικό περιθώριο με το σενάριο της μιας μέρας χωρίς συμψηφισμό και επίσης στη συνέχεια για δύο μέρες με συμψηφισμό. Αυτά τα στοιχεία βασίστηκαν σε πραγματικά στοιχεία που συλλέγουμε ως τμήμα της εποπτείας της Επιτροπής μας. Και τα δώσαν τα στοιχεία αυτά στην Κομισιόν. Τα στοιχεία αυτά αφορούν επτά μέρες ε, εργάσιμες. Βλέπετε ότι με την ε, διαδικασία της μιας μέρας χωρίς συμπληρωματισμό φτάνουμε στα 58 δισεκατομμύρια συνολικό περιθώριο, ενώ με το σύστημα δύο ημερών με συμπληρωματισμό με του ίδιου αντισυμβαλόμενου θα φτάναμε μονάχα στα 23 δισεκατομμύρια περιθώριο. Η διαφορά είναι 35 δισεκατομμύρια δολάρια σε αρχικό περιθώριο το οποίο πρέπει να έχει ο κεντρικός αντισυμβαλόμενο. Περίπου 150% διαφορά και περαιτέρω. Έτσι η ανάλυση μας από τα εννέα μεγαλύτερα κεντρικά αποθετήρια οδηγούν, σε, όπως είπα, σε περίπου 1,6 με 4 φορές περισσότερο στη διαδικασία που δεν έχει συμψηφισμό. Ας δούμε τώρα το περιθώριο το οποίο οφείλει ο κεντρικός αντισυμβαλόμενος, το οποίο δεν μπορεί να συγχέεται με το περιθώριο που πρέπει να καταθέσουν οι συμβαλόμενοι. Εδώ, για δύο μέρες με συμψηφισμό, έχουμε περισσότερα ποσά από ότι για μία μέρα, και εδώ φυσικά αυτό μπορεί να το περιμένει κανείς γιατί δεν υπάρχει συμψηφισμός. Μιλάμε για τον κεντρικό αντισυμβαλόμενο και τη θέση που έχει έναντι των, ε, των πελατών. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει πάλι διαφορά του 41% που ανέφερα προηγουμένως. Αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι η συνολική θέση του κεντρικού αντισυμβαλωμένου στις αγορές προθεσμιακών συμβολέων είναι πολύ μικρότερο ποσό από το συνολικό ποσό για το σύνολο των, επι... των Επομένως, το περιθώριο είναι της τάξης του 14% ίσως και τόσο λίγο όσο 10% εναντί του συνολικού περιθωρίου των ε, συμβαλωμένων. Έχουμε λοιπόν στον, στο γράφημα 4 το απαιτούμενο περιθώριο με πραγματικά στοιχεία Σήμερα έχουμε 9 δισεκατομμύρια. Αν ακολουθούσαμε το ευρωπαϊκό σύστημα, αυτό θα αύξανε το περιθώριο σε 13 δισεκατομμύρια ενάντια 9. Αλλά υπάρχει και μια περαιτέρω διαφορά ότι αν αντιμετωπίσουμε τους, ε, τους ε, φορείς οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με τον κεντρικό ε, αντισυμβαλόμενο που ε, συνδέονται, που καταλογίζονται μάλλον στον κεντρικό λογαριασμό του κεντρικού αντισυμβαλωμένου και όχι ως πελάτες. Επομένως, με την λογική αυτή, το δεύτερο τμήμα του γραφήματος 4 δείχνει τι θα γινόταν αν ακολουθούσαμε ευρωπαϊκούς κανόνες. Η διαφορά λοιπόν ανάμεσα στο συνολικό περιθώριο του κεντρικού αντισυμβαλωμένου εάν δεν λάβουμε υπόψη τους συνδεόμενους με τον κεντρικό λογαριασμό τότε θα είχαμε 3,6 δισεκατομμύρια για μία μέρα και 5,1 δισεκατομμύρια για δύο μέρες. Πάλι η διαφορά είναι περίπου 1,5 δισεκατομμύρια. Το πέμπτο γράφημα σας δείχνει τον αντίκτυπο του δικού μας ρυθμιστικού πλαισίου με τα πραγματικά στοιχεία που ανέφερα. Στην κορυφή λοιπόν του γραφήματος 5 βλέπετε τη διαφορά όπως τη βλέπει ο πελάτης. Τα 58 δισεκατομμύρια είναι αυτά που πρέπει να καταθέσουν οι συμβαλόμενοι έναντι 23 δισεκατομμύριων, ενώ το κάτω διάγραμμα δείχνει το περιθώριο του ίδιου του κεντρικού αντισυμβαλωμένου χωρίς τους συνδεόμενους χωρίς που θα είναι 3,6 δισεκατομμύρια έναντι 5,1. Μιλάμε λοιπόν για μια διαφορά που είναι πολύ μεγαλύτερη, 35 δισεκατομμύρια από την πλευρά των πελατών, έναντι μιας διαφοράς που θα είναι για τον κεντρικό αντισυμβαλόμενο μόνο 1,5 δισεκατομμύρια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα έχει την ε, ε, ανησυχία ότι το μικρότερο περιθώριο για τον κεντρικό αντισυμβαλόμενο μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί κίνδυνο. Δεν υπάρχει λοιπόν λέει μεγαλύτερο κίνδυνο αθέτηση από τον κεντρικό αντισυμβαλόμενο. Βεβαίω υπάρχει μικρότερο περιθώριο, αλλά η μεγάλη, μεγαλύτερη απειλή είναι η διαφορά σε συνολικό περιθώριο για τους, για τους ε, Εάν υπάρξει αθέτηση από το κεντρικό της συμβαλόμενο, το θέμα είναι πώς θα προστατεύσουμε τους συμβαλωμένους και πώς θα πρέπει να αποτρέψουμε το να χρειαστούν τα, οι άλλοι κεντρικοί αντισυμβαλόμενοι να πληρώσουν τη διαφορά. Το συνολικό περιθώριο για τους συμβαλόμενους είναι αυτό το οποίο θα προσδιορίσει το κατά πόσο οι πελάτες αυτού του κεντρικού αντισυμβαλόμενου μπορούν να μεταφερθούν σε κάποιο άλλο κεντρικό συμβαλόμενο ή αν θα πρέπει να εκαθαριστούν οι θέσεις τους, κάτι το οποίο οδηγεί σε ε, ανασφάλεια και αστάθεια στις αγορές. Είναι αντίστοιχο με την περίπτωση της Lehman Brothers. Αν μπορούμε λοιπόν με τη μεταφορά να μειώσουμε τις ανάγκες σε εγγύησεις. Και αυτό εξασφαλίζει το ότι θα είναι μικρότερη η εμπλοκή του Ταμείου Εγγύησεων. Έτσι λοιπόν, Εάν πράγματι θέλουμε εμείς να μιλήσουμε γενικότερα για χρηματοπιστωτική σταθερότητα, έχουμε να κερδίσουμε περισσότερα μέσω της συνολικού υπολογισμού παρά της αύξησης της ελάχιστης περίοδου πληρωμής στους εσωτερικούς λογαριασμούς ενός ε, αντισυμβολωμένου. Γιατί θα μου πείτε. Γενικά βλέπουμε ότι οι, Αμερικανοί, οι αμερικανικές εταιρείες αντισυμβαλόμενοι χρησιμοποιούν είτε μία, περίοδο, μία περίοδο μίας ημέρας είτε ε, μία περίοδο δύο ημερών. Η περίοδος πληρωμής αποφασίζεται ανάλογα με το προϊόν και ανάλογα με τα ε, χαρακτηριστικά κινδύνου του συγκεκριμένου προϊόντος. Για κάποια προϊόντα είναι μία μέρα, για άλλα προϊόντα είναι περισσότερο. Για τα swaps θα έπρεπε να είναι και πρέπει να είναι, συμφωνούμε όλοι πέντε μέρες. Και ανησυχούμε γιατί ε, η διαφορετική περίοδος υπολογισμού ανάλογα με το ποιος κατακρατά το προϊόν θα δημιουργήσει κίνητρα για να ξεφύγει κανείς από τον κανονισμό και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλουμε να ξεφύγουμε, δηλαδή το διακανονιστικό αρμπιτράζ, τη διακανονιστική διαιτησία. Θα είναι ιδιαίτερα προβληματικό αυτό εάν η Ευρώπη και οι Ηνωμένε Πολιτείε χρησιμοποιούν και αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο τις θηγατρικές εταιρείε ή τις εξαρτημένες εταιρείε. Στις Ηνωμένε Πολιτείε, σαν παράδειγμα, θα προσπαθήσουν να εμφανιστούν σαν πελάτες στην Ευρώπη για να ξεφύγουν ακριβώς τους αμερικανικούς κανονισμούς. Και σίγουρα το περιθώριο είναι κάτι το σχετικό με μια στάση πληρωμών. Και αυτό το οποίο επίσης παίζει ρόλο είναι η συνεισφορά του Ταμείου Εγγυήσεων. Και το ποσό από τη μία πλευρά είναι κάτι που θα επηρεάσει αν πολύ στο ποσό και της άλλης πλευράς. Είπα στην αρχή ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να τα αντιμετωπίσει όλα αυτά κανείς συνολικά, ολιστικά και να δούμε και άλλους κινδύνους και τρόπους μείωσης των κινδύνων. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αξιολογήσουμε ε, και το, τη συνολική εικόνα ενός νομικού και εποπτικού πλαισίου. Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές στα πλαίσια μας. Σε κάποιους τομείς οι ευρωπαϊκοί κανόνες είναι πολύ πιο συντηρητικοί. Και υπάρχουν άλλοι τομείς στους οποίους οι δικοί μας ε, κανόνες είναι πολύ πιο συντηρητικοί, δεσμευτικοί. Θα το συζητήσουμε αυτό αν θέλετε. Ο στόχος μας να πρέπει να δούμε ποιος είναι. Προσπαθούμε να εξισώσουμε τις διαφορές μας. Θέλουμε να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στην, στην χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Εάν ναι, τότε θα πρέπει να ξεκινήσουμε με το περιθώριο του πελάτη. Εκεί υπάρχουν οι μεγάλες διαφορές. Θα πρέπει να δούμε ακριβώς ποια είναι τα συναλλικά ποσά, ποια είναι η υποχρεωτική συλλογή των περιθωρίων αυτών για τους πελάτες. Αυτές είναι οι διαφορές οι οποίες εφόσον ε, ξεπεραστούν θα βελτιώσουν την ε, χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την προστασία του πελάτη. Και η σωστή τοποθέτηση, η συνολική τοποθέτηση των θέσεων του πελάτη είναι κάτι το οποίο έτσι κι αλλιώ ελέγχεται σε άλλες δικαιοδοσίες ε, και δικαιοδοσίες τις οποίες έχουμε ήδη χορηγήσει την αντιστοιχία που απαιτείται. Πρέπει να συνδυάσουμε τις διαφορές λοιπόν, όπως επίσης και τις διαφορές στην αντιμετώπιση των συνδεδεμένων εταιριών ή των θηγατρικών. Και εκεί είναι ένας άλλος τρόπος για να βγάλει χρήματα ένα μέλος ενός clearing house, ενός αποθετηρίου. Μαζί με τη συνεισφορά του Ταμείου Εγγυήσεων, αν δούμε ότι όλα αυτά δεν είναι επαρκή σε περίπτωση στάσης πληρωμών, τότε θα πρέπει να προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε. Αλλά θα πρέπει να αποφύγουμε να δημιουργήσουμε κίνητρα τα οποία θα οδηγήσουν σε ε, συμπεριφορές αποφυγής του διακανονιστικού πλαισίου και σε σχέση με την περίοδο ε, πληρωμής. Όλα αυτά είναι αρκετά τεχνικά βέβαια τα οποία σας είπα, λυπάμαι γι' αυτό, αλλά ελπίζω να σας βοήθησαν έτσι ώστε να μπορέσετε να συνειδητοποιήσετε ακριβώς ότι έχουμε μπροστά μας, τι πρέπει να συζητήσουμε. Είμαι στη διάθεσή σας να δώσω απαντήσεις πάνω σε αυτά τα οποία σας είπα ή και να συζητήσουμε θέματα παραγόγων ή άλλα θέματα τα οποία έχετε στην, στο νου Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Thank you. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μάσαντ για την παρουσίασή σας η οποία ήταν πάρα πολύ τεχνική. Αλλά καταλαβαίνετε καλύτερα τα τεχνικά στοιχεία. Άλλο η σαφήνεια, άλλο η συμφωνία. Και τώρα θα πρέπει να ακούσουμε τα μέλη της Επιτροπής μας. Φυσικά θα ε, υποβληθούν διάφορες ερωτήσεις, μεταξύ των οποίων ε, και εγώ θα σας κάνω ερωτήσεις. Θεωρείτε σημαντικό ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν λογαριασμοί των ε, πελατών για να καλύψουν τις απώλειες εντός του γραφείου συμψηφισμού και τι εννοείται όταν λέτε ότι θα πρέπει να δούμε να δούμε τους τρόπους για να αλλάξουμε αυτό το στοιχείο. Στο τελευταίο σημείο της ομιλίας σας το αναφέρατε. Το βασικό θέμα της διαφορετικής μεταχείρισης για τους ε, εσωτερικούς λογαριασμούς ε, είναι με ποιο τρόπο μπορούμε να αλλάξουμε αυτές τις διαφορές, να εξομαλύνουμε αυτές τις διαφορές. Δεν, δεν νομίζω ότι η Επιτροπή αυτή είναι η πιο αρμόδια για την εξασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Ε, η Επιτροπή λέει για τη σημασία ε, των εσωτερικών λογαριασμών σε αντιδιαστολή με, τον, με τους ε, λογαριασμούς των πελατών. Αυτές είναι οι πρώτες ε, ερωτήσεις. Ε, Βεβαίω να σας απαντήσω. Πιστεύουμε στεναρά ότι τα λεφτά των πελατών δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν τις την πτώχευση σε περίπτωση του γραφείου, ας πούμε, συμψηφισμού ή του κεντρικού αποθετηρίου. Ε, γι' αυτό απαιτούμε από τους συνδεδεμένους, ε, αν η Goldman Sachs, ας πούμε, είναι τέτοιο μέλος, δεν πιστεύουμε ότι... US, ε, Goldman Sachs, ε, είναι μέλος, δεν πιστεύουμε ότι η Goldman Sachs International πρέπει να είναι ε, εντός του... Τα λεφτά της πρέπει να συνυπολογίζονται εντός του γραφείου αυτού συμψηφισμού. Εσεί είπατε ότι εγώ θέλω να το αλλάξουμε αυτό. Όχι, δεν θέλω να αλλάξουμε αυτό τον διαχωρισμό. Αυτή η διαχωριστική γραμμή πρέπει να υπάρχει. Είναι σημαντικό νομίζω να αναγνωρίσουμε ότι αν υπάρχει πτώχευση στο γραφείο συμψηφισμού, ε, προφανώς θα έχουμε και θέματα και προβλήματα με τους λογαριασμού των πελατών το μέγεθος της έκθεσης είναι πολύ μεγαλύτερο και τα θέματα είναι πολύ μεγαλύτερα όταν πίν η Λίμαν ή οποιοδήποτε τέτοια εταιρεία πτωχεύει. Ανησυχούμε για το τι θα γίνει με τους πελάτες. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει πτώχευση, το μέλος ε, του γραφείου δεν θέλει να πληρώσει τίποτα. Γιατί φοβάται τι θα γίνει με την ε, διαμάχη και τι θα γίνει με τη διαδικασία αφαιρεκιότητας, τα πάντα παγώνουν. Και το Γραφείο Συμψηφισμού θα πρέπει να αποφασίσει εάν θα μεταφέρει αυτού του λογαριασμού αν μπορεί, των πελατών. Αυτό θα εξαρτηθεί από το περιθώριο που υπάρχει. Μια άλλη εταιρεία μπορεί να μην αναλάβει τι θέσει αυτέ των πελατών, εάν δεν υπάρχει επαρκέ περιθώριο. Γι' αυτό λοιπόν συμφωνώ ότι πρέπει να ανησυχούμε για το τι συμβαίνει ε, με τους λογαριασμού αυτούς του εσωτερικούς, αλλά αν υπάρχει πτώχευση, θα τεθούν θέματα για το λογαριασμό των πελατών, τους λογαριασμού των πελατών. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πόσα λεφτά έχουν αυτοί οι λογαριασμοί των πελατών. Με ρωτήσατε τι πιστεύω για μια τέτοια αλλαγή. Δεν μιλάω για κατάρριξη του διαχωρισμού αυτού. Πιστεύουμε ότι τα πράγματα αυτά δεν πρέπει να ανακατευτούν. Τι εννοούσα, ότι αν τα λεφτά τους εσωτερικούς λογαριασμούς δεν αρκούν, θα πρέπει να ψάξουμε να δούμε τι εγγύσει υπάρχουν. Γιατί και εκεί βάζουμε χρήματα τα μέλη ε, του Γραφείου Ψηφισμού. Θα πρέπει να δούμε το, το κεφάλαιό τους. Και θα πρέπει όλα αυτά να τα δούμε μαζί και να αποφασίσουμε αν αρκούν αυτά τα λεφτά. Ε, μην ξεχνάμε όμως ότι μιλάμε για κάποια ποσά εδώ. Τα λεφτά, τα εσωτερικά, ε, είναι πολύ λιγότερα από τα λεφτά των πελατών. Είναι σημαντικό. Δεν λέω ότι δεν είναι. Αλλά υπάρχει εδώ ο ελέφαντας που είναι τα λεφτά των πελατών και υπάρχει κάτι πολύ μικρότερο που είναι τα λεφτά του γραφείου συμψηφισμού. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ασχολούμαστε και με τα δύο και είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ευχαριστώ. Αν είναι τόσο μικρό το ποσό, γιατί έχετε δυσκολία να το αυξήσετε, βέβαια, λέει ο πρόεδρο Γουαλτιέ. Μα δεν θέλουμε να το αυξήσουμε μόναχα με το να πάμε στις δύο μέρες και έχουμε άλλη μια μέρα για το λογαριασμό του πελάτη. Αυτό θα δημιουργήσει ακριβώς τον κίνδυνο ε, ρυθμιστικού αρμπιτράς, δηλαδή επιλογής ρυθμιστή. Κύριε Μπουκαμπάλτση, η οποία είναι συντονιστή. Α, ο κύριος Μπάλτση, συγγνώμη. Ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε Μασάτ. Σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας σήμερα. Είναι πολύ καλό που έχετε έρθει στις Βρυξέλλες. Εμείς στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων γνωρίζουμε πολύ καλά ποια είναι η σημασία του, της συνεργασίας μεταξύ των δύο οχτών του Ατλαντικού σε ό,τι αφορά τα θέματα της χρηματοπιστητικής ρύθμισης. Θα ήθελα λοιπόν και πάλι να έρθω σε ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα που φυσικά θα συζητηθεί και από άλλους ε, ομιλητές σήμερα που είναι ακριβώς αυτό το περιθώριο που απαιτείται για λόγους ασφαλείας στα κεντρικά αποθετήρια. Εμείς στην Ευρώπη θέλουμε να εξασφαλίσουμε την σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών. Αυτό είναι το κύριο μας εγχείρημα, κύρια μας μέρημνα. Γι' αυτό θα ήθελα να σας θέσω το ερώτημα. Ε, το εξής. Πρώτα απ' όλα το ερώτημα κατά πόσον θα ήταν πιο πιθανό ένα κεντρικό αποθετήριο έχει να αντιμετωπίσει ε, μια ανάγκη αθέτησης πληρωμών για κάποιον ο οποίος είναι συνδεόμενος με το κεντρικό αποθετήριο από ότι με ένα πελάτη. Και το δεύτερο πρόβλημα, το δεύτερο ερώτημα που ήδη έχετε αναφέρει εν μέρη, αλλά θα ήθελα να το ξαναθέσω για να σας δώσω τη δυνατότητα να μας δώσετε περισσότερα στοιχεία ενδεχομένω. το θέμα του υψηλότερου περιθωρίου ασφαλείας που θα, τον, από την πλευρά των πελατών που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εξίσωση οφειλών προς τους ε, συνδεόμενους με το κεντρικό ε, αποθετήριο. Πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό αν δεν έχουμε υψηλότερα περιθώρια ή αν δεν έχουμε τη δυνατότητα πληρωμής σε δύο μέρες. Θα ήθελα λοιπόν να εξηγήσετε τη θέση σας για αυτό το θέμα, εάν μπορείτε. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα προσπαθώ να ε, εξασφαλίσω ότι κατάλαβα το ερώτημά σας γιατί δεν φόρησα τα ακουστικά μου όταν ξεκινήσατε το, την παρέμβασή σας. Πρώτον είναι ρωτήσατε αν το ίδιο το κεντρικό αποθετήριο, ο κεντρικό αντισυμβαλόμενο δεν έχει μεγαλύτερη πιθανότητα αθέτησης πληρωμών. Και δεύτερον, αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, μήπω πρέπει να απαιτήσουμε υψηλότερο περιθώριο για τον κεντρικό αντισυμβαλόμενο. Σε ό,τι αφορά την πιθανότητα αφέτηση πληρωμών, η δική μα άποψη είναι ότι αν έχετε μία αθέτηση από το κεντρικό αντισυμβαλόμενο, δεν είναι μονάχα θέμα των λογαριασμών αυτού του κεντρικού αποθετηρίου. Θα πρέπει να δει κανείς συνδυασμένα και τους λογαριασμούς των πελατών και του κεντρικού αποθέτη. Και λόγω της σχέσης μεταξύ των δύο, του σχετικού μεγέθους, ο κίνδυνος για, τον, το κεντρικό αντισυμβαλόμενο και τα άλλα συμβαλόμενα μέρη προέρχεται κυρίως από το αν έχει επαρκές περιθώριο ο λογαριασμός των πελατών. Σκεφτείτε εδώ πόσο μεγάλες είναι οι διαφορές. Οι διαφορές μεταξύ 35 δισεκατομμυρίων για τους πελάτες και αυτό είναι περίπου 4 δισεκατομμύρια για κάθε μία από τις 9 εταιρείες που εμπλέκονται. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποιο είναι το... η αναλογία σε αυτή την περίπτωση. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να μας απασχολήσει και το περιθώριο ασφαλείας που έχει και το κεντρικό αποθετήριο, ο κεντρικό αντισυμβαλόμενο. Αυτό φυσικά είναι ένα σημαντικό θέμα, <clears throat> αλλά εκεί θα πρέπει να εξετάσουμε το σύνολο των μέτρων και των διαδικασιών που έχουμε για να αποτρέψουμε την αφαίρεση πληρωμών από την πλευρά του κεντρικού αντισυμβαλωμένου και το πώ θα αντιμετωπίσουμε αυτή την περίπτωση. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη και το Ταμείο Εγγυήσεων, τα χρήματα τα οποία δίδονται για το Ταμείο Εγγυήσεων, όπου συμβάλλουν τα κεντρικά αποθετήρια και που είναι το δεύτερο τείχο, το δεύτερο ανάχωμα κατά κάποιο τρόπο σε περίπτωση αθλέτησης πληρωμών. Γι' αυτό πρέπει εμείς να παρακολουθούμε όλα αυτά, κάνουμε κάθε μέρα μετρήσεις για να ξέρουμε πόσο μεγάλη είναι η έκθεση των κεντρικών αποθετηρίων. Η δική μου λοιπόν ανησυχία αν αντιμετωπίσουμε το θέμα λέγοντας μία μέρα εδώ, δύο μέρες εκεί. Δημιουργεί αυτό ε, κίνητρα για μία συμπεριφορά η οποία προσπαθεί να αποφύγει στη ρύθμιση. Προσπαθούν κάποιοι να κάνουν ε, συναλλαγές ως πελάτες, ενώ ουσιαστικά αυτό το κάνουν ως κεντρικοί αντισυμβαλόμενοι. Γιατί λέμε λοιπόν ότι χρειάζεται περισσότερο περιθώριο από την πλευρά του κεντρικού αντισυμβαλωμένου και αν θεωρείται θεωρείτε ότι αρχή αρκετό, ας προσπαθήσουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και εδώ νομίζω ότι πρέπει να δείτε ακριβώς ποια είναι η συμβολή και η εμπλοκή του Ταμείου Εγγύησεων. Γιατί είναι το περιθώριο συν τις συνεισφορές στο Ταμείο Εγγύησεων που είναι το συνολικό ποσό που ουσιαστικά επιτρέπει να υπάρχει πλήρη κάλυψη. Ίσως θα πρέπει να δούμε πώς ε, μετράμε αυτό το ποσό, το λεγόμενο cover to, το, το συνολικό ποσό που είναι το περιθώριο συν το Ταμείο Εγγύησεων. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να μην είναι αρκετό αυτό το ποσό του cover του, του ποσού αυτού του συνολικού. Εμείς λέμε απλώς όμως ας προσπαθήσουμε, εάν θεωρούμε, να, θεωρούμε ότι δεν επαρκείς η, η ασφάλεια από το περιθώριο του κεντρικού αντισυμβαλωμένου υπάρχουν άλλοι τρόποι να αντιμετωπίσουμε αυτό το, το, το, το θέμα και όχι να έχουμε αυτή τη διαφορά μεταξύ των δύο του Ατλαντικού που θα οδηγήσει σε ρυθμιστικό αρμπιτράζ. Ο Φενάντε Αλβάρε έχει το λόγο από του σοσιαλιστέ. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε. Κύριε Μασάντ, είναι μια μεγάλη τιμή να μπορούμε να σας υποδεχτούμε στην Επιτροπή μας. Και μεταξύ άλλων θα έχουμε αυτή την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτό το θέμα που φαντάζομαι ότι αυτό σας έφερε στις Βρυξέλλες για να προσπαθήσετε να επιλύσετε τις διαφορές στη διαπραγμάτευση για τα περιθώρια των κεντρικών αντισυμβαλωμένων και των πελατών τους. Ένα από τα διδάγματα που έχουμε αποκομίσει από την χρηματοπιστωτική κρίση είναι ότι δεν αρκεί να μειώνουμε τον μεμονωμένο κίνδυνο κάθε οικονομικού παίκτη στην κανονική του δραστηριότητα, υπάρχει και ένας συστημικός κίνδυνος, κάτι που για πάρα πολλά χρόνια έχει εκφύγει από την ανάλυση των ρυθμιστικών αρχών και των υποπτών ακόμα και η ακαδημαϊκοί μελετητέ δεν το είχαν λάβει υπόψη αυτόν τον συστημικό κίνδυνο και αυτός λοιπόν ο κίνδυνος θα πρέπει να, να ληφθεί υπόψη στη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Γι' αυτό η Βασιλεία 3 για τους τραπεζικού φορείς περιλαμβάνει πρόσθετα μέτρα ελέγχου για να ελέγξει όχι μόνο τον ατομικό κίνδυνο κάθε τράπεζα ή κάθε οικονομικού φορέα, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτή η, η, η δραστηριότητα μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους που διαχέονται στο σύνολο του συστήματος και επομένως πρέπει να αντιμετωπιστούν. Λαμβάνοντα τώρα υπόψη τις διαφορές στα ρυθμιστικά συστήματα των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής έχει κανείς την εντύπωση ότι το αμερικανικό σύστημα κατά πάσα έχει και ένα περιθώριο για τους πελάτες, απαιτούμενο περιθώριο για τους πελάτες που είναι υπέρτερο αυτού που απαιτείται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αντίθετα όμως, το περιθώριο για τον κεντρικό αντισυμβαλόμενο φαίνεται να είναι μεγαλύτερο βάσει των στοιχείων που έχει η Κομισιόν όχι των δικών σας στοιχείων, αλλά των στοιχείων μας έχει δώσει η Κομισιόν από την ευρωπαϊκή πλευρά. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει κάπως μεγαλύτερη έμφαση στο συστημικό κίνδυνο με το γεγονός ότι το περιθώριο για τον κεντρικό αντισυμβαλόμενο περιλαμβάνει ε, και κάποιο αποθεματικό για αυτόν τον κίνδυνο που δεν έχουν οι λογαριασμοί των πελατών. Για να μπορέσουμε όμως να αποφύγουμε αυτό το ρυθμιστικό αρμπιτράζ, την επιλογή μεταξύ των δύο δικαιοδοσιών, που μπορεί να οδηγήσει αμερικανικές εταιρείες, να, ευρωπαϊκές εταιρείες να λειτουργούν στις ΗΠΑ, θα ήθελα να σας ρωτήσω γιατί εσείς δεν δέχεστε το να υπάρχουν δύο ημέρες για το διάστημα πληρωμής χωρίς συμψηφισμό, ώστε να υπάρξει μια συμβαστική λύση μεταξύ της ευρωπαϊκής και της αμερικανικής λύσης σε ποιο βαθμό δεν θα είχαμε μεγαλύτερη συστημική προστασία με το να έχουμε μεγαλύτερο αποθεματικό ασφαλείας στον, ε, στο αμερικανικό σύστημα αντισυμβαλωμένο, γιατί να μην έχουμε ένα πιο ελαφρό σύστημα με αυτό το σύστημα των δύο ημερών χωρίς συμπληκτισμό. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι βασικός μας στόχος είναι να αντιμετωπίσουμε τις πιθανότητες συστημικού κινδύνου. Μάθαμε πολλά από την κρίση. Μάθαμε ότι μπορεί να υπάρξει μια σόρευση υπερβολικών κινδύνων σε ορισμένε αγορές που δεν είχαμε συνειδητοποιήσει ότι υπήρχαν και υπήρξε η χώρα μου χρειάστηκε πέντε χρόνια για να βγει από αυτό. Και θα συμφωνήσω λοιπόν με τα σχόλιά σας. Να μην ξεχνάμε όμως αυτά τα οποία μάθαμε στην κρίση. Γενικά ε, τα περιθώρια για τις προθεσμιακές συναλλαγές δεν είχαν καμία σχέση, δεν προκάλεσαν την κρίση. Τα παράγωγα ήταν σχετικά και ιδιαίτερα τα εντελώς αρρύθμιστα θα λέγαμε, μη, εποπτευόμενα τέτοια παράγωγα. Um, Αυτά τα οποία ήσαν εκτός αγοράς. και εκεί υπήρξαν κάποιες συζητήσεις και είπαμε μέχρι σε ποιο επίπεδο οι διαφορές θα ήσαν αποδεκτές. Το μεγαλύτερο, το σημαντικότερο θέμα για μένα, για, για, τον, για τον κίνδυνο αυτό, δεν έχει καμία σχέση με τις προθεσμιακές συναλλαγές, αλλά έχει να κάνει με τα swaps τα οποία δεν έχουν περάσει από τα αποθετήρια. Μιλάμε για ένα μεγάλο τμήμα της αγοράς το οποίο δεν περνά από τα αποθετήρια σε καμία περίπτωση. Και εμείς και εσείς προσπαθούμε να βρούμε κάποιους κανόνες ως προς αυτό. Εμείς προτείνουμε ένα πολύ χαμηλότερο επίπεδο ε, περιθώριο σχετικά με, το, με την πρόταση την οποία είχαμε κάνει και την οποία απέρριψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άλλωστε. Εγώ είπα πάντως ότι είμαι διατεθειμένος να ακολουθήσω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν και θα προτιμούσαμε ένα χαμηλότερο ποσοστό. Θα προτιμούσαμε κάτι το οποίο θα μας παρέχει, νομίζουμε, καλύτερη προστασία. Αλλά παρόλα αυτά, αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους και το κόστος της εποπτείας αυτής, του διακανονισμού αυτού τη ρευστότητα των αγορών αυτών. Αυτές οι αγορές είναι εξαιρετικά ωφέλιμες για τις οικονομίες μας και τις επιχειρήσεις και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη. Και εγώ συναντώ εκπροσώπους γενικά των αγορών οι οποίοι δεν έχουν καμία ε, σχέση με τους συστημικούς κινδύνους επαφίενται στις αγορές αυτές για τα προϊόντα τους και για τα γεωργικά προϊόντα και για τις, για τις βιομηχανικές δραστηριότητες και για τις εξαγωγικές δραστηριότητες για να καλύψουν τους κινδύνους τους νομισματικούς. Και αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε με ποιο τρόπο δεν πρέπει να επηρεάσουμε αρνητικά το κόστος των προϊόντων τους, των αγαθών τους. Πιστεύουμε λοιπόν ότι οι μεθοδολογίες του περιθωρίου που ακολουθούμε σήμερα που οδηγούν στη μία μέρα για τα περισσότερα από αυτά τα συμβόλαια είναι κατάλληλες ρυθμίσεις και δεν είχαμε προβλήματα στην κρίση με αυτό. Υπάρχουν βέβαια πολλές παρατηρήσεις και πολλά ενδιάμεσα, δεν είναι από τη μία μία μέρα και από την άλλη δύο μέρες. Συζητήσαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ιδανική σε σχέση με τη διαμόρφωση του κινδύνου, πώς αντιμετωπίζει ε, κανείς ε, το θέμα του χρόνου γενικότερα και την προκυκλικότητα. Η ανησυχία μου λοιπόν είναι ότι ξαφνικά συγκεντρώνουμε την προσοχή μας σε ένα θέμα το οποίο θα το έλεγα δευτερεύον. Ενώ υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά θέματα τα οποία θα πρέπει να τεθούν σε συζήτηση και μιλάμε ε, για τις διαφορές στον εσωτερικό λογαριασμό του αποθετηρίου για ε, αν θα υπάρξει μία μέρα ή δύο μέρες. Ε, το θέμα είναι σημαντικό, αλλά υπάρχουν πολύ σημαντικότερα θέματα. Και δεύτερον, υπάρχουν και άλλες πολιτικές και άλλες ρυθμίσεις και διαδικασίες οι οποίες επηρεάζουν αυτό το καθεστώς στο σύνολό του. Τρίτον, εφόσον κάνουμε τις αλλαγές τις οποίες ζητάτε, ε, θα δημιουργήσουμε πολύ περισσότερη διακανονιστική διαιτησία την οποία θα θέλαμε να αποφύγουμε. Στόχος μας αυτός είναι. Λοιπόν θα ήθελα να ζητήσω παρακαλώ τους ομιλητές να μην ξεπερνούν το πεντάλεπτο ο καθένας. Γι' αυτό οι ερωτήσεις σας παρακαλώ πολύ επαναλαμβάνω να είναι σύντομες. Και η απάντηση πρέπει να είναι σε ένα πεντάλεπτο. Στάνισλαβ Χοζόκ από το ECR. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκ μέρου τη ε, συναδέλφου μου, τη κυρία Σουίνβερτ, η οποία δυστυχώ δεν μπορούσε να παραστεί σήμερα, η ερώτησή μου αφορά την ισοδυναμία. Δεν θα σε εκπλήξει. Δεδομένων των διαφορών που υπάρχουν ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην ε, Επιτροπή Προθεσμιακών Συμβολέων Επιαγαθών. Το να βασιζόμαστε περισσότερο σε διεθνή πρότυπα για να μετρήσουμε το αποτέλεσμα νομίζουμε θα οδηγήσει σε λιγότερες προστριβές μεταξύ των διαφορών περιοχών του πλανήτη. Πρόσφατα ακούσαμε μία δήλωση της Επιτροπής σας που είπατε Ε, για τη δουλειά που κάνει τη δουλειά η Όσκο, που λέει ότι δεν δεσμεύονται ε, σε ό,τι αφορά τις εξουσίες που έχουν. Και θέλουν περισσότερους λεπτομερείς κανόνες σε διεθνές επίπεδο σε ό,τι αφορά τα πρότυπα για τα περιθώρια, ε, τα stress test και την δυνατότητα ανάκαμψης των CCP. Αυτό θα κάνει το πλαίσιο πολύ πιο διαφανές και θα υπάρχει μεγαλύτερη λογοδοσία. Και με αυτόν τον τρόπο δεν θα γίνουν μικρότερες οι διαφορές μεταξύ των διαφορετικών δικαιοδοσιών και δεν θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για το θέμα της ισοδυναμίας. Ε, και θα, θα έχουμε λιγότερες διαφορές, οποίες θα πρέπει να ξεπεράσουμε. Ευχαριστώ για την ερώτησή σα. Για την αίσθηση, για την υποσημείωση αυτή που αναφέρατε. Να σας πω ποιο είναι το πλαίσιο. Ο λόγος που ζήτησε κάτι τέτοιο το SEC και που το υποστηρίξαμε είναι η φύση των νομικών και κανονιστικών μας υποχρεώσεων. Και εκείνο και εγώ είμαστε πρόεδροι επιτροπών. Η Επιτροπή μπορεί να δράσει μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια και Επιτροπή Κεφαλαίου επίσης. Ναι. Εμείς οτιδήποτε αποφασίσουμε θα πρέπει να το υποβάλουμε στην Επιτροπή Κεφαλαίου Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι μόνοι μας. Εγώ υποστηρίζω την δουλειά που κάνει η Όσκο αυτή τη στιγμή. Ε, τα stress test, το θέμα της ε, ε, διάλυσης και της Και εμείς και εσείς έχουμε κανόνες, νομοθεσία και βεβαίως και οι διεθνείς διαδικασίες είναι πολύ σημαντικές ε, για να θέσουμε κάποια πρότυπα. Το κάναμε για τα περιθώρια. Έχουμε τα PFMI που είναι κανόνες ε, σημαντικοί Τώρα, αν θα πρέπει να γίνουμε πιο λεπτομέρειες στους κανόνες μας. Θα ήταν δύσκολο να ξαναρχίσουμε λεπτομερείς συζητήσει για τα μάρτζινα, για τα περιθώρια. Αλλά βεβαίως εγώ υποστήριζω τη δουλειά που γίνεται σε άλλους τομείς. Υπάρχουν θέματα που έχουμε να συζητήσουμε διμερώς ακόμα. Νομίζω ότι είναι στοιχείο της δουλειάς μας αυτό, στοιχείο του τομέα μας εγγενές στοιχείο. Ευχαριστώ. Η κόρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε Μασάντ, που βρήκα το χρόνο και κάνα την προσπάθεια να έρθετε εδώ για να ανταλλάξουμε απόψεις, όπου, σε ένα κόσμο όπου οι κεφαλαγορέ είναι όλο και πιο συνδεδεμένε και είναι σημαντικό οι χώρε και οι διάφορε δικαιοδοσίε να έχουν συνεχή διάλογο για να έχουν νομοθεσίε οι οποίες λειτουργούν Ισχύει αυτό και για τον προτινόμενο κανονισμό για τα benchmark, όπου είμαι εισηγήτρια. Και η μεταχείριση των, εξω, των μη Ευρωπαίων παραγωγών ήταν σημαντική. Από την αρχή της νομοθετικής διαδικασίας στην Επιτροπή είχαμε συνεχείς διαδικασίες, ε, συζητήσεις με εποπτικές αρχές και με ρυθμιστικές αρχές από όλες τις χώρες, Σιγκαπούρη, Ιαπωνία, Ινδονησία, ε, Νότια Αφρική. Όλες αυτές οι χώρες και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εκφράσει ανησυχίες ό,τι αφορά το καθεστώ των τρίτων χωρών, όπως είχε προταθεί αρχικά. Τα benchmarks που υπάρχουν σε άλλα τμήματα του κόσμου χρησιμοποιούνται από τους Ευρωπαίους επενδυτές και καταναλωτές σε καθημερινή βάση και σε ό,τι αφορά τα μη ευρωπαϊκά benchmark, εγώ εστίασα σε τρία στοιχεία. Πρώτον, έχουμε την υποχρέωση να εξασφαλίσουμε ότι χρησιμοποιούμε τα πρότυπα με στεναρό τρόπο και ότι δεν υπάρχει καμία κατάχρηση ή λαθροχειρία. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα benchmark των τρίτων χωρών πρέπει να χρησιμοποιούνται από τι τράπεζε σε επενδυτέ ε, επιχειρήσει και νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτον, θα πρέπει να δημιουργήσουμε ε, ισοτιμία για τα ευρωπαϊκά ε, benchmark και οι Ευρωπαίοι και οι μη Ευρωπαίοι συμβαλόμενοι να αντιμετωπίζονται επί συσσόρισης. Εσείς καθαρίσατε ότι το CFTC και όλοι οι άλλοι φορείς δεν έχουν ε, εντολή για να εποπτεύσουν τους, τους φορείς των benchmark. Πρόσφατα είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να θεωρήσει το αμερικανικό καθεστώς ε, ισοδύναμο με της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί ε, έμεσα υπάρχει μέσω του delisting και της εποπτείας έλεγχος στα benchmark. Θα μπορούσατε να μας δώσετε παραδείγματα του CFTC που χρησιμοποιεί τις εξουσίες delisting είτε μέσω της απειλής απλώς. Η CFTC θέλει ε, τα διάφορα γραφεία να συμμορφούνται με τις αρχές IOSCO. Θα χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα να διώξει από το χρηματιστήριο οποιοδήποτε φορείς προκειμένου να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις αρχές ΙΟΣΚΟ. Ελπίζω να συμφωνείτε ότι δεν θα πρέπει να γίνει μια μάχη ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη δική σας Επιτροπή για το ποιο έχει το πιο αυστηρό σύστημα, για το ποιος κανονισμός είναι καλύτερο, γιατί όπως είπαν και οι συνάδελφοι, Παίζονται πάρα πολλά. Και τα γραφεία συμψηφισμού είναι πολύ σημαντικά για όλο το σύστημα. Να σα ρωτήσω και αυτό, ξανά αυτό που σα ρώτησα στην από την ECR. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε κοινά α, νέα πρότυπα σε διεθνέ επίπεδο. Ίσως θα μπορούσαμε να το πετύχουμε μέσω τη IOSCO ή με άλλο τρόπο. Σα ευχαριστώ για το ερώτημα. ο τρόπος με τον οποίο έχουμε αντιμετωπίσει το θέμα των benchmarks είναι ο εξή. Όπως είπατε, έχουμε μια διαδικασία εποπτείας όπου ένα νέο συμβόλαιο στην αγορά μελλοντική εκπλήρωσης θα πρέπει να τύχει επαναθεώρησης από εμά και βλέπουμε αν βασίζεται σε κάποιο βασικό επιτόκιο, παραδείγματος σε κάποιο benchmark, θεωρούμε αν μπορεί να υφίσταται κίνδυνος ε, χειραγώγησης ή απάτης. Εγώ θα χαιρόμουν πάρα πολύ. Δεν μπορώ τώρα αυθόρμητα να σας δώσω κάποιο ιστορικό παράδειγμα. Είχαμε τα... <laughs> το παράδειγμα του bitcoin που μας οδήγησε σε κάποιες ανησυχίες πρόσφατα. <clears throat> Αλλά έχουμε κάνει κάποιες προσπάθειες να τροποποιήσουμε ακόμα και τρέχοντα συμβόλαια εάν ε, θεωρούσαμε ότι δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε να λειτουργήσουν. Περαιτέρω όμως δεν είναι μονάχα η επιθεώρηση των συμβολέων, αλλά είναι και η διαδικασία εφαρμογής. Όλες οι περιπτώσεις του Libor το 2012 ήρθαν στην επιφάνεια από εμά. Και ξεκινήσαμε μια δικαστική διαδικασία μαζί με την αρχή χρηματοπιστωτικών αγορών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Deutsche Bank χρειάστηκε να, κατα... να καταβάλει πρόστιμα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν λοιπόν όλες αυτές οι κυρώσεις, υπάρχουν όλες αυτές οι απαιτήσει που προκύπτουν από τη διαδικασία της ε, χειραγώγησης του LIBOR, του, της διατραπεζικής ε, μέρα ε, αγοράς μιας μέρας από το Λονδίνο. Όλα αυτά λοιπόν βασίζονται στις ίδιες αρχές όπως οι αρχές της ΙΟΣΚΟ. Δεν κάνουμε ε, κάποια επίσημη ρύθμιση για τα βασικά επιτόκια. Αυτό το ξέρετε, δεν μπορούμε λοιπόν, τα επιτόκια αναφοράς, δεν μπορούμε λοιπόν να υποχρεώσουμε όλους να ακολουθούν τις αρχές του, της Ιόσκο. Χρησιμοποιούμε όμως αυτά τα πρότυπα, παρόμοια πρότυπα της Ιόσκο, στην δική μας δράση. Τα χρησιμοποίησαμε για τα επιτόκια αναφοράς όπως της Λίμπορ, για τα για τις ισοτιμίες που ισχύουν για τις αγορές, προθεσμιακές αγορές συναλλάγματος κτλ. Είναι λοιπόν στοιχεία τα οποία εμπίπτουν στη διαδικασία μας ε, ε, εποπτείας και εφαρμογής κανόνων. Όπως ξέρετε είχαμε εμπλακεί ιδιαίτερα στην διατύπωση των αρχών της ΙΟΣΚΟ. Έχουμε συμβάλει πάρα πολύ σε αυτή τη διαδικασία και οι φορείς οι οποίοι μας δίνουν αναφορές σε σχέση με τις τιμές της αγοράς, όχι μοναχά παρακολουθούν τις αρχές της ΙΟΣΚΟ για τις τιμές πετρελαίου που ήταν το αντικείμενο της έκθεσης της ΙΟΣΚΟ που αναφέρατε, αλλά έχουν μεταφέρει αυτή τη μεθοδολογία και σε άλλους δείκτες τιμών. Είναι διαφορετικό σύστημα λοιπόν. Δεν έχουμε μια επίσημη διακυβέρνηση για τα επιτόκια αναφοράς ή τους δείκτες αναφοράς, αλλά μας ενδιαφέρει να εξασφαλίσουμε την ακαιρεότητα αυτών των δικτών αναφοράς και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξασφαλίσουμε ότι αυτοί οι δείκτες δεν υπόκεινται σε χειραγώγηση ή σε απατηλές ε, συναλλαγές. Ελπίζω ότι έχω απαντήσει το ερώτημά σας. Ευχαριστώ. Για την ομάδα της ΓΚΟΕ, ο Φάβιο Δημάσιο. Ευχαριστώ κύριε Μασάτ για τον χρόνο που μας δίνετε. Θέλω να σταθώ στο όριο των θέσεων στις αγορές βασικών προϊόντων. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες και υπάρχει η ανάγκη αναφορών, αλλά από ό,τι γνωρίζω ανεστάλησαν μετά από μια δικαστική απόφαση που είπε ότι η Αμερικανική κυβέρνηση δεν είχε καταδείξει την αναγκαιότητα αυτών των κανόνων για να περιστήλουν την κερδοσκοπία και από ό,τι ξέρω η CFTC προσπαθεί τώρα να αναθεωρήσει αυτούς τους κανόνες και περιμένει ότι αυτό θα γίνει μέχρι το τέλο του 2015. Νομίζω ότι από αυτό μπορούμε να βγάλουμε κάποια διδάγματα για το πώς θα πρέπει να σχεδιάσουμε του δικού μα κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μην έχουμε τα ίδια προβλήματα. Θα ήθελα όμως να σα ρωτήσω το εξή. Ποια είναι η δική σα κρίση για τις εξελίξει που έχουν αυξήσει τα όρια για την απόδοση αναφορών σε σχέση με τις ε, θέσεις που υπάρχουν ε, των ε, εμπορευμένο σε ένα συγκεκριμένο χώρο και όταν μιλάμε τώρα πάλι για τα κεντρικά αποθετήρια, τους κεντρικούς αντισυμβαλωμένους. Όταν μας λένε, όταν τους ρωτάμε για, τις, ε, για τα παράγωγα της τράπεζας, λένε δεν έχουν σημασία οι θέσεις μας, έχουν σημασία μόνο οι καθαρές μας θέσεις μετά από συμπλησφισμό. Εσείς λέτε ότι η προτού, η έκθεση προτού συμψηφισμού είναι πιο καλό μέτρο κινδύνου. Εσείς θεωρείτε ότι οι θέσεις χωρίς συμψηφισμό δίνουν μια καλύτερη εικόνα του εγγενούς κινδύνου που αντιμετωπίζει ένας κεντρικός αντισυμβαλόμενος και αν μου επιτρέψει τώρα και ο πρόεδρος ή θα σας επιτρέψει να απαντήσετε μάλλον υπήρξε μια πρόσφατη περίπτωση με, ένα, με σύλληψη ενός ε, συμβαλόμενου σε χρηματιστήριο που χρησιμοποίησε τη μέθοδο της υψηλής συχνότητας και οδήγησε σε χρηματιστηριακό κράχ θα ήθελα και εγώ να εκφράσω την ε, απορία μου για το αν ένας μονάχα εμπορευόμενος μπορεί να οδηγήσει σε τόσο μεγάλη κατάρρευση και θα ήθελα να ξέρω ποια είναι δική σας άποψη για το θέμα αυτό. Για τα όρια θέσεων. Εμείς προσπαθούμε να φτάσουμε σε αναφερεμένους κανόνες. Ακυρώθηκε από το δικαστήριο ένας κανόνας, ή μάλλον ένας κανόνας που είχε προταθεί πριν από τρία χρόνια ίσως κάτι τέτοιο. Είναι τεχνικό διαδικαστικό το θέμα. Δεν είναι θέμα αυστήρα νομικό. Βέβαια η εντολή την οποία πήραμε εμείς από το Κογκρέσο ήταν συγκεκριμένη να καταθέσουμε εκ νέου ένα κανόνα θα το κάνουμε αυτό, το προετοιμάζουμε και ελπίζουμε μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουμε προχωρήσει. Σε σχέση με τα υπόλοιπα, δεν είμαι εμπειρογνώμων στα όρια αυτά και δεν μπορώ να τα σχολιάσω. Ελπίζω όμως ότι μπορούμε να συντονιστούμε. Είναι κάτι το αρκετά δύσκολο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσπαθήσουμε για, το, για τα παράγωγα. Μιλάμε για τους αντισυμβαλόμενους, μιλάμε για τις πολιτικές των τομέα των, των ορίων. οι τράπεζες μερικές φορές παραπονούνται για, τις, για την έκθεσή τους. Ίσως να μην κατάλαβα καλά αυτό που είπατε, αλλά το θέμα δεν αρκεί κανείς να βλέπει ακριβώς την ε, συνολική έκθεση σε μια δεδομένη στιγμή. Η απάντηση που θα μπορούσε κανείς να δώσει είναι ότι περνάμε σε, ένα είδος συλλογικότερης αντιμετώπισης του προβλήματος του χρέους. Δεν ξέραμε ακριβώς το τι γινόταν σε επίπεδο έκθεσης. Στην ουσία ήταν ένας από τους λόγους που έστειλε τις οικονομίες μας στην ύφεση. Αυτό το οποίο πρέπει να προσπαθήσουμε τώρα είναι να υπολογίσουμε την έκθεση και την καθαρή έκθεση των τραπεζών σαν παράδειγμα, αλλά και των συσχετισμών που δημιουργούνται. Ε, τι σημαίνει η έκθεση ενός μεγάλου ε, οικονομικού ιδρύματος σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται με ένα άλλο μικρότερο. Όλοι κατανοούμε ότι τα swaps είναι προϊόντα τα οποία μερικές φορές μπορεί να είναι ενός είδους ε, πιο επικίνδυνο από ό,τι, άλλα, από κάποιο άλλο. Αλλά όλα αυτά απαιτούνται να υπολογιστούν για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε σωστά το εύρος της έκθεσης για την τελευταία σας παρατήρηση ερώτηση. Ευχαριστούμε εδώ και την συνεργασία και της FCA και της Scotland Yard εμείς ε, προχωρήσαμε σε αστική και ποινική δίωξη εναντίον ενός ε, χρηματιστή από τις Ηνωμένε Πολιτείες στην Ευρώπη. Εμείς αυτό το οποίο είπαμε και αυτό το οποίο πιστεύουμε είναι ότι αυτού του είδους οι συμπεριφορές οδήγησαν στην δημιουργία κάποιων συνθήκων στην αγορά που στην ουσία οδήγησαν στο λεγόμενο flash clash. και υπάρχει ένα συγκεκριμένο προϊόν, εν το οποίο ε, χρησιμοποιήθηκε. Ακολούθησε κάποιες στρατηγικές, οι οποίες στην ουσία ε, δημιουργούσαν οι στρατηγικές αυτές μια διατεταγμένη αταξία θα το έλεγα αυτή, έτσι ώστε να καταφέρει να ρίξει την τιμή του προϊόντος τους. Το flash crash ήταν συνδυασμός πολλών ε, υποθέσεων. σχετικά τώρα με τις αυτοματοποιημένες ε, μορφές ε, χρηματιστηριακών συναλλαγών. Έχουμε κάνει διάφορα προς την κατεύθυνση αυτή από το flash crash και προσπαθούμε ε, να δούμε τώρα ποιος είναι ο πραγματικός κίνδυνος για τις αγορές μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Μασάτ που ήρθατε να μας απαντήσει σε ερωτήσεις. Ε, η ερώτηση μου είναι ανάλογη με αυτή που έκανε ο συνάδελφός μου από την ΚΟΕ όπως και ο συνάδελφος από την ECR ε, και εγώ ε, εκφράζω τις απόψεις κάποιου άλλου συναδέλφου για ε, τα όρια των θέσεων. Είπατε ότι δεν έχετε πολλές λεπτομέρειες για αυτά που προτείνουμε, αλλά ε, αυτό το όριο των 40% ε, ορισμένοι είπαν ότι είναι πολύ ψηλό για να οδηγήσει σε στρέβλωση της αγοράς γιατί τρεις φορεί θα μπορούσαν να ελέγξουν την αγορά χωρίς να σπάσουν τα όρια. Τώρα κάτι δικό μου όμως, για τη διαπραγμάτευση των παραγών, παραγωγών επί βασικών αγαθών όπως τροφίμων ας πούμε. Εσείς έχετε αρκετή εμπειρία. Ε, για μένα και για τους πολίτες είναι ε, προβληματικό να σκέφτομαι ότι κάποιοι κερδοσκοπούν ε, πάνω σε βασικά αγαθά όπω τα τρόφιμα. Ε, και ορισμένοι αντισταθμίζουν το κίνδυνό τους ούτως ώστε να εξασφαλίζονται απέναντι σε διακοιμάσεις στην αγορά. Τι φιλοσοφική άποψη έχετε για τα τρόφιμα και τα βασικά άγαθα που θεωρούνται ε, περιουσιακά στοιχεία, στοιχεία του ενεργητικού. Τι γίνεται με τη διαπραγμάτευση σε τέτοιου τύπου ε, αγαθά που έχουν υποτίθεται κοινωνική αξία, κοινωνική λειτουργία και όχι και δεν θα πρέπει να έχουν κερδοσκοπική ας πούμε, ε, λειτουργία. Αυτό που εγώ σκέφτομαι είναι, συνδέεται με το τι σκέφτομαι για τα όρια των θέσεων. Υπάρχει χώρος για μια κερδοσκοπία, για μια κάποια κερδοσκοπία, αλλά θέλουμε να αποφύγουμε την υπερβολική κερδοσκοπία. Και το θέμα είναι η οριοθέτηση που θα κάνουμε. Υπάρχει χώρος για κερδοσκοπία. Ο αγρότης ο οποίος να προσπαθεί να αντισταθμίσει τον κίνδυνο για διακύμανση ας πούμε, των τιμών του αραβοσίτου, ας πούμε, Εμείς ε, αυτούς που αγοράζουν ας πούμε, τα παράγωγα τους θεωρούμε κερδοσκόπους γιατί δεν ασχολούνται οι ίδιοι με γεωργικά προϊόντα, δεν είναι οι ίδιοι γεωργοί ας πούμε. Χωρίς αυτούς όμως ο, ο γεωργός δεν μπορεί να αντιμετωπίζει τον πιθανό κίνδυνο ας πούμε της τιμής και ίσω μπορεί να μην καλλιεργήσει και ποτέ. Τι κάνουμε εμεί λοιπόν με τον κανόνα για τα όρια θέσεων. Είναι να αποφύγουμε την υπερβολική κερδοσκοπία που μπορεί να επηρεάσει την διαθεσιμότητα αυτών των αγαθών τελικά, αυτών των βασικών προϊόντων. Σε ό,τι αφορά το 40% είναι υψηλότερο από αυτό που προτείναμε εμεί, Άρα υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία σε αυτούς του κανόνες και φυσικά υπάρχουν άτομα στο γραφείο μου που ξέρουν πολύ καλύτερα από όλα αυτά τα στοιχεία. Εγώ δεν είμαι εμπειρογνώμονας. Δεν είμαι τεχνικός. Πρέπει να κοιτάξετε και τα όρια. Είτε μιλάμε για στιγμή αγορά, για spot market ή όχι, για υπερβολική έκθεση, θα πρέπει ε, να δούμε σε τι βασίζουμε τον υπολογισμό των ε, παραγόγων. Ε, υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που επισέρχονται για να δούμε πού θα, κάνουμε, θα βάλουμε αυτή τη διαχωριστική γραμμή. Εμείς όλα αυτά τα παίρνουμε όλα αυτά πολύ σημαντικά. Εμείς ξεκινήσαμε στην Επιτροπή μου από τη Γεωργία. Επομένως, είμαστε ακόμα και τώρα εστιασμένοι στα γεωργικά θέματα και προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι οι γεωργοί στη χώρα μας και καταλαβαίνω ε, ότι όταν λέμε γεωργοί, μερικέ φορέ εννοούμε και μεγάλε γεωργικέ εκμεταλλεύσει. Αλλά τέλο πάντων η παραγωγή τροφίμων για τι οικογένειέ μα να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν αυτέ τι αγορέ αποτελεσματικά. Αυτό. Ε, κοιτάξτε, ε, εμείς μιλάμε για την εμπορική σημασία αυτών των αγοράων. Ε, και όχι, θα πρέπει να εξυπηρετούν αυτή την ε, εμπορική ας πούμε, λειτουργία και όχι να προωθούν την κερδοσκοπία των χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Αυτή είναι η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε καθώς προσπαθούμε να διαμορφώσουμε αυτούς τους κανόνες. Ευχαριστώ. Από την EFTD, ο Μάρκο Βάλλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μασάντ που ήρθε εδώ και που μας παρουσίασε την τεχνική αυτή θέση που ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Χαίρομαι που υπάρχει αυτή η διάθεση συνεργασίας γιατί καταλαβαίνουμε το συστημικό κίνδυνο που υπάρχει. Και θέλουμε φυσικά να τον διασκεδάσουμε αυτόν τον κίνδυνο. Ε, θέλουμε να, έχουμε, να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα ε, παγκόσμια. Για την ισοδυναμία με τις ΗΠΑ έχουμε σοβαρές αμφιβολίες, ακούστηκαν ήδη και από άλλους για το θέμα της ε, εξισορρόπησης ε, του συμψηφισμού. Φυσικά υπάρχουν κάποια στοιχεία υπέρ της δικής μας ε, θέσης και κάποιες φορές υπέρ της δικής σας. Ακούμε επικρίσεις. Κατά εμά θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια για αυτά τα εργαλεία για να μην υπάρχει κερδοσκοπία στι πρώτε ύλε, ε, στα κρατικά ομόλογα, όπου υπήρχαν περιπτώσει και στην Ιταλία προβληματικέ με υπερβολική κερδοσκοπία, να μην τι εξηγήσω τώρα. Και για τα swap επίση προσπαθήσαμε να προστατευτούμε κάπως. Τελικά χρειάστηκε να πληρώσουμε πολύ περισσότερο. Ε, από, υπήρξε μια μείωση των επιτοκίων, αλλά τελικά χρειάστηκε να πληρώσουμε πολύ, πιο, πολύ περισσότερο από ό,τι περιμέναμε. Τι άποψη έχετε για το να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός φερμός ε, θεσμός στην Ευρώπη ε, όπως ο δικός Αμερικάνικος που κάθε τρεις μήνες ε, ε, δημοσιεύει τις θέσεις των πιο σημαντικών Αμερικανικών τραπεζών. Εμείς έχουμε πάρα πολύ χονδροειδείς, ας πούμε, εκτιμήσεις ε, για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, για τις μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες. Θα θέλαμε συγκεκριμένα στοιχεία. Έχει νόημα να δημιουργήσουμε και εμείς έναν ευρωπαϊκό, ας πούμε, φορέα που θα κάνει αποτίμηση των, ευρωπαϊκών, των μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζών. Συμφωνώ ότι χρειαζόμαστε καλύτερη κατανόηση και μεγαλύτερη ακρίβεια στα θέματα αυτά. Είναι πολλά πράγματα όμω τα οποία γίνονται προ την κατεύθυνση αυτή. Βέβαια δεν είμαι εγώ αρμόδιο να σχολιάσω τα, του, τα θεσμικά όργανα που χρειάζεται η Ευρώπη για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά. Όλοι όμω εμπλεκόμαστε στη διαδικασία αυτή που αφορά την οικοδόμηση ενός συστήματος για την ε, ε, συλλογή και δημοσίευση δεδομένων για τα παράγωγα μέσα από τα κεντρικά αποθετήρια. Και εμείς έχουμε ξεκινήσει, έχουμε εγκρίνει νομοθεσία και εσείς έχετε ζητήσει υποχρεωτικά να γίνονται αναφορές σε σχέση με τις συναλλαγές σε swaps. Αυτό λοιπόν το οποίο προσπαθούμε να οικοδομήσουμε θα είναι ένα πολύ καλύτερο σύστημα, πολύ πιο λεπτομεριακά, πολύ πιο πληροφοριακό σύστημα από ό,τι το OCC, το Office of the Control of the Currency, κάνει σήμερα. Γίνονται πολλές προσπάθειες να εναρμονιστεί αυτό. Μιλάμε πολύ για την εναρμόνιση. Νομίζω ότι προχωρούμε σημαντικά σε ό,τι αφορά την, ε, ε τις αναφορές για τα swaps. Πιστεύω λοιπόν ότι μαζί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, εμείς έχουμε συμπροεδρεύσει στη συνολική αυτή προσπάθεια. Όπως λοιπόν προχωρούμε για τη δημιουργία αυτού του συστήματος, αυτό θα οδηγήσει σε καλύτερα στοιχεία για την αγορά αυτή, οπότε θα μπορούμε να δούμε πού βρίσκονται οι εκθέσεις, πού βρίσκονται οι κίνδυνοι. Έχουμε βέβαια ακόμα δυσκολίες για να επιμεριζόμαστε τα δεδομένα, να, για να εναρμονίσουμε επίσης τα πρότυπά μας, νομίζω ότι γίνονται θετικές προσπάθειες για τα θέματα αυτά. Κατά πόσο η Ευρώπη πέραν αυτό χρειάζεται να οικοδομήσει κάποια άλλα εργαλεία, αυτό είναι κάτι που εσεί πρέπει να κρίνετε και όχι εγώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Από ό,τι ξέρω, έχετε ακόμα 8 λεπτά. Ίσως μπορούμε να ομαδοποιήσουμε τα τελευταία ερωτήματα. Για... Η Μπάρμαρα Κάπελ για τους μη εγγεγραμμένους. Ένα λεπτό, ένα μισή λεπτό το πόλι παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Μασάρ για την τόσο ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας για την Αμερικανική μεθοδολογία που έχει να κάνει και με τα θέματα της ε, ε, αμοιβαία αναγνώσης και ισοδυναμίας των κεντρικών αντισυμβαλωμένων. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα γενικά για τα παράγωγα και τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών. Σε μία συνεδρίαση των G20 υπήρξαν κάποιες βασικές αρχές που διατυπώθηκαν για τα εκτός αγοράς παράγωγα. Θεωρήθηκε ότι πρέπει να γίνονται η ε, εμπορία όλων των swaps σε οργανωμένες αγορές και μέσω κεντρικών αποθετηρίων. Αυτά θεωρήθηκαν από ότι είναι μια μορφή προστατευτισμού. Εσείς έχετε ζητήσει να γίνεται η, η ανταλλαγή swaps, η εμπορία swaps μέσω κεντρικών αποθετηρίων για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος. Στις ΗΠΑ βέβαια υπάρχουν οι μεγαλύτερες αγορές παραγόγων και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα πολύ μικρότερο ποσό τέτοιων ε, ε, παραγόγων και η Ευρώπη διδάσκεται πολλά από τα δικά σας συστήματα. Θα ήθελα να δω από τη δική σας άποψη η ευρωπαϊκή νομοθεσία με το MIFID για την ε, ε, αγορά, για τα εκτός αγοράς παράγωγα έχει χαρακτήρα προστατευτισμού και πώς βλέπετε τους ρυθμιστικούς στόχους στην Ευρώπη έναντι αυτών των Ηνωμένων Πολιτειών. Πώς αντιμετωπίζετε τη MIFID και πού βλέπετε να υπάρχουν οι διαφορές μεταξύ της νομοθεσίας Dot Frank στις ΗΠΑ και της ε, οδηγίας MIFID στην Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των παραγωγών. Πάρα πολλά ερωτήματα λέει ο πρόεδρος, ο Brian Hayes. Πάρα πολύ σύντομα κύριε πρόεδρε και εγώ καταλαβαίνω ότι ο κύριος Μασάτ πρέπει να φύγει. Είσαστε ιδιαίτερα καλόδεκτο στην Επιτροπή σα. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπατε σε σχέση με τα όρια θέσεων, σε σχέση με τα παράγωγα. Αυτό είναι ένα θέμα που αντιμετωπίζουμε τώρα στα πλαίσια τη MIFID και προσπαθούμε να βρούμε και κάποιο τρόπο να βελτιώσουμε την νομοθεσία στον τομέα αυτό. Έχω ένα συγκεκριμένο ερώτημα για σα μονάχα. Είναι σωστό το να πω ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν την άποψη ότι παρά το γεγονό η, η ΟΣΚΟ θέτει διεθνεί αρχέ και πρότυπα. Οι Ηνωμένε δεν θέλουν μια ρυθμίση που να είναι οικουμενική για όλο τον κόσμο παρά το γεγονό ότι έχουμε προχωρήσει πολύ από το 2008, εσεί είχατε το Federal Reserve και μπορέσατε να λύσετε την κρίση πιο εύκολα. Εμεί χρειάστηκε να φτιάξουμε τα τεστ αντοχή, να φτιάξουμε το CRD4, τη διαδικασία επίλυση και ανάκτηση. Είναι λογικό να πούμε ότι καταρχήν η Ιόσκα, η Ιόσκο συμφωνεί για πρότυπα, αλλά μετά κάθε περιοχή, κάθε χώρα θα πρέπει να εφαρμόσει αυτά τα πρότυπα με τον δικό τη τρόπο. Αυτό επαρκεί κατά τη δική σα άποψη λόγω τη κλίμακα των προβλημάτων που εξακολουθούν να υφίστανται. Πάρα πολύ σύντομα. Ο κύριο Φερνάντε, αν είσαστε. Σύντομα, κύριε Φερνάντε, παρακαλώ. Και μετά θα δώσω το λόγο στην Επιτροπή και σε εσάς κάτι το πολύ συγκεκριμένο. Θα ήθελα να μάθω το θέμα της συμπερίληψης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στο εσωτερικό του DTIP, τη Συμφωνία της Εμπορικής με τις ΗΠΑ. Θα ήθελα να μάθω ποια είναι η άποψή σας και ποια είναι η άποψη επίσης πάνω στο θέμα το οποίο προσπαθούμε εμείς να κάνουμε εδώ, να ελέγξουμε δηλαδή με πιο λεπτομερή τρόπο τη συμφωνία αυτή, ε, και επίσης ε, και τον ρόλο τον οποίο και την άποψή σας για τον ρόλο τον οποίο μπορεί να παίξουν ε, οι, τα συνδικάτα. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Μασάντ, ευχαριστώ και το προσωπικό. Το Συμβούλιο έδωσε μια συγκεκριμένη εντολή να προχωρήσει σε συμφωνίες αντιστοιχίας με συγκεκριμένες χώρες. Ε, θα πρέπει ακριβώς να υπάρξει αναφορά λοιπόν στους κανόνες μας σε συγκεκριμένη χώρα και θα συμφωνήσω με τα σχόλια του Τιμ Μασάντο ότι στα πλαίσια της συζήτησης που έγινε με τις ΗΠΑ υπήρξαν σημαντικά βήματα πρόοδου. Οι κανόνες για τρίτες χώρες θα πρέπει να είναι αντίστοιχοι, ομόλογοι με τους δικούς μας. Αυτό δεν είναι κάτι το καινούριο εδώ και πάρα πολύ καιρό και στο, στην ιστοσελίδα της CFTC e είχαμε στείλει μια επιστολή λέγοντας ότι είχαμε ανησυχίες σε σχέση με τα περιθώρια αυτά των πελατών. Γιατί έχουμε. Γιατί η ΑΙΟΣΚΟ έχει υιοθετήσει κάποια διεθνή standards, αλλά υπήρχαν κάποιοι τομείς τους οποίους δεν θα μπορούσαν να συμφωνήσουν και ήταν τα περιθώρια. Τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητούσαν ε, να υπάρξει εναρμόνιση, αλλά υπήρχαν και κάποιες διαφοροποιήσεις μεταξύ μας. Και αυτό ήταν ένα πρόβλημα. Αν υιοθετήσουμε μία απόφαση για αντιστοιχεία, ευρωπαϊκά CCP που θέλουν να μπουν στην Αμερικανική αγορά θα πρέπει έτσι και αλλιώς να σεβαστούν ε, τις αντίστοιχες ε, ρυθμίσεις της Αμερικανικής αγοράς οι ε, αντισυμβαλόμενοι οι Ευρωπαίοι χρησιμοποιούν όταν παρεμβαίνουν στις αμερικανικές αγορές ε, τους κανόνες οι οποίοι ισχύουν στη ΣΥΠΑ. Τώρα θα πρέπει να επιτρέψουμε εμείς σε αμερικανικούς τέτοιους οίκους ε, αντίστοιχα να παρεμβαίνουν στις δικές μας αγορές. Αυτό είναι το ερώτημα και ο κύριος Φερνάντες, ο κύριος Μπάλτς και άλλοι είπαν ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα. Στην Ευρώπη το θέμα που απασχολεί το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο είναι η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Το περιθώριο δηλαδή των αντισυμβαλωμένων απέναντι στα επιμέρους μέλη τους. Οι μεγάλες τράπεζες, Barclays, ε, JP Morgan, Deutsche Bank, Goldman Sachs. Εκεί θέλουμε να υπάρχουν οι δυνατότητες αποζημιώσεων. Εκεί βρίσκεται η σταθερότητα, η σταθεροποίηση της αγοράς. Εκεί θα προστατεύσουμε σωστά τους πελάτες. Αυτό είναι το θέμα για μας. Υπάρχουν λοιπόν περιθώρια βελτίωσης στην, στις Ηνωμένε Πολιτείε. Στην Ευρώπη έχουμε κάποια υψηλότερα επίπεδα προστασίας. Το θέμα είναι πώς θα τα όλα αυτά. Δεν θα πρέπει απλά να δεχθούμε την πρόταση η οποία λέει ότι θα πρέπει να υπάρξουν υψηλότεροι αριθμοί στις ΗΠΑ, πελατών και χαμηλότερη τέχη ε, στην Ευρώπη γιατί δεν μπορεί να υπάρξει μια απλή ανταλλαγή. Ακόμα χειρότερα, αν μια πολύ μεγάλη τράπεζα συμπαρασύρει τους αντισυμβαλωμένους σε μια στάση πληρωμών και αν πράγματι δημιουργηθεί μια τέτοια καταστροφή τότε το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έχουν κάνει μια συγκεκριμένη επιλογή. Θα πρέπει εμείς να προχωρήσουμε στην προστασία των CCP, των αντισυμβαλωμένων απέναντι στις μεγάλες ε, εταιρείες. Πραγματικά εδώ έχουμε βγει να διαφημίζει ο καθένας ε, ποιανού οι κανόνες είναι καλύτεροι. Πρέπει να υπάρξει μια αντιστοιχία και δεν θα πρέπει να λέει μια τέτοια επιχείρηση αντισυμβαλωμένων στην ε, Ευρώπη ότι θα πρέπει να μεταναστεύσει στις Ηνωμένε Πολιτείες για να έχει πιο συμφέρουσες ρυθμίσεις. Πώς μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε. Είναι αρκετά θέματα τεχνικά. Έτσι κι αλλιώς σκεφτόμαστε μια αύξηση του περιθωρίου. Θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί σας περαιτέρω και ο Μασάντ και οι συνάδελφοί του συνεχίζουν να εξετάζουν τα θέματα αυτά. Θέλουμε να προχωρήσουμε στην εναρμόνιση των περιθωρίων και στα πλαίσια της ΑΙΟΣΚΟ, κάτι το οποίο δεν πετύχαμε εδώ και κάποια χρόνια. Οι αγορές όμως απαιτούν μεγαλύτερη ευκρίνεια. Δεν μπορούμε εμείς ε, συνεχώς να παρατείνουμε τους ισχύοντες κανόνες. Απαιτείται μια βραχυπρόθεσμη λύση. Και ελπίζω και στη συνάντηση του Μασάντ με τον Επίτροπο Χίλ αύριο να υπάρξει αυτή η συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μασάντα, έχει το λόγο. Να απαντήσω. Και τα θέματα διαπραγμάτευσης. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε τη δουλειά μας πιο ενεργά. Να κοιτάξουμε δηλαδή πώς εναρμόσουμε τους ε, κανόνες διαπραγμάτευσης ακόμα περισσότερο. Είναι σημαντικό να το κάνουμε. Δεν θέλω να μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες, γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Ένα-δύο πράγματα θα να πω. Ε, το, Κόγκρε, το Κογκρέσο μας ζήτησε να εφαρμόσουμε τους κανόνες μας στην Ευρώπη. Γι' αυτό κινήθηκε γρήγορα η υπηρεσία μας. Είναι δύσκολο προφανώς όταν έχεις ε, μια παγκόσμια αγορά που δεν ήταν καθόλου ρυθμισμένη. Καμία χώρα δεν είχε προβεί σε κανονιστική ρύθμιση. Ε, μια χώρα, ας πούμε, έχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο διαπραγμάτευσης ε, όταν το δημιουργήσει πριν από τις υπόλοιπες χώρες, τότε δημιουργούνται προβλήματα. Ε, περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει η Ευρώπη και προσπαθούμε να εναρμονίσουμε τους κανόνες όσο μπορούμε. Το μόνο που θέλω να πω είναι για το θέμα της εναρμόνισης. Ειλικρινά σας το λέω, ότι κάνουμε πολλά για να εναρμονίσουμε. Ο κλάδος ε, ε έρχεται και μου λέει ότι οι κανόνες ε, εναρμον, εναρμονίζονται υπερβολικά. Γιατί γιατί είναι συνηθισμένοι στο να μην υπάρχουν καθόλου κανόνε. Είναι μεγάλη αγορά επίση. Θα εναρμονίσουμε όσο μπορούμε. Ίσως υπάρχουν μικρέ διαφορέ, ούτω ε, ή άλλω υπάρχουν πολλέ διαφορέ και ο κλάδο μπορεί να τους αντιμετωπίσει. Εγώ ασχολούμαι με, με τις κινητές αξίες πολλά χρόνια. Δεν μπορεί να πουλήσετε ε, κινητές αξίες με τον ίδιο τρόπο α πούμε, στην Ευρώπη και στην Αμερική και στην Ιαπωνία κτλ και προσαρμόζεται ο κλάδο κάθε φορά. Εναρμονίζουμε όσο μπορούμε, στο βαθμό που μπορούμε, αλλά α μην μα πιέσουν για να φτάσουμε στην απόλυτη εναρμόνιση, ότι πρέπει να υπάρχει απόλυτη συνέπεια και σαφήνεια. Είναι θαυμάσιο ο σκοπό, είναι φιλοδοξία, αλλά είναι δύσκολο να υλοποιηθεί. Δεύτερον, η βασική αρχή στη χώρα μα είναι ότι σεβόμαστε την νομοθεσία μας. Πιστεύουμε στεναρά στην διαδικασία της ΙΟΣΚΟ. Ε, συζητούμε τις διεθνείς συζητήσεις, τη διεθνή συνεργασία, την FSB, παρότι δεν είμαι μέλος. Χαίρομαι που βλέπω ότι υπάρχει. Τα πρότυπα που, προ, που προκύπτουν από τις διεθνείς διαδικασίες ε, επειδή δεν είμαστε ένα πράγμα, δεν υπάρχει ένας παγκόσμιος, μια παγκόσμια εθνιστική αρχή, εμείς ως χώρα θα αποφασίσουμε αν θα εφαρμόσουμε ή όχι. Αρκούν. Τι να κάνουμε, αυτά έχουμε. Πρέπει να κάνουμε ότι μπορούμε το καλύτερο. Ε, θα μπει στο TTP, στο TTIP οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Δεν είναι θέμα της αρμοδιότητάς μου. Ε, όλα τα... Το πλαίσιο που έχουμε μας εξυπηρετεί νομίζω καλά. Το μόνο που μπορώ να πω αναφέρθηκε κάτι σε συνδικάτα, το οποίο δεν το κατάλαβα. Μπορείτε να με ρωτήσετε μετά για να σας απαντήσω. Και τώρα, για τα σχόλια του Πάτρικ Τίρσον, Η ιδέα ότι οι κεντρικοί αδεσυμβαλόμενοι ε, θα πρέπει να σέβονται όλους τους Αμερικανικούς κανόνες για να κάνουν δουλειά στην Ευρώπη δεν είναι αλήθεια. Εμείς δεν εμποδίζουμε τους Αμερικανούς να διαπραγματεύονται προθεσμιακά συμβόλαια στην Ευρώπη. Και μπορούμε να τα... Δεν εμποδίζουμε κανέναν Ευρωπαίο αντισυμβαλόμενο, ας πούμε, να ασχολείται με προθεσμιακά συμβόλαια οποιασδήποτε φύσεως. Ούτε swaps. Το ευρωπαϊκό καθεστώς είναι διαφορετικό. Θα επιβάλλεται ε, επιβαρύνσεις ε, σε οποιονδήποτε αντισυμβαλόμενο που δεν αναγνωρίζετε εσείς στην Ευρώπη. Εμείς δεν έχουμε πιο καθεστώς. Η υποχρέωσή μας για την καταχώρηση ενός αντισυμβαλόμενου είναι πολύ πιο χαλαρή από αυτή που περίεψε ο Πάτρικ. Η ιδέα επίσης ότι δεν ενδιαφερόμαστε για τις μεγάλες τράπεζες και τις, τους κινδύνους που δημιουργούν στο σύστημα δεν ισχύει, δεν είναι σωστό. Και ελπίζω να μην χρειάζεται να το συζητήσουμε αυτό με μεγάλη χαρά να συζητήσω όλους τους τρόπους που παρακολουθούμε τα μέλη των ε, γραφείων συμψηφισμού και προστατεύουμε εναντίον των περιπτώσεων ε, θέτησης ε, της υποχρέωσης πληρωμής κτλ. Γι' αυτό λέω, ας μην εστιάζουμε σε μία μονοπτυχία, σε εξασφαλίσουμε ότι έχουμε μία συνολική θεώρηση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι μας ανησυχεί και εμάς, όπως και εσάς, ο κίνδυνος που θέτουν ε, οι μεγάλοι, τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο σύστημα. Το σχόλιο μου για τα όσοι είπες Πάτρικ είναι ότι οποιαδήποτε στοιχεία μας δώσεις να τα δούμε, να τα εξετάσουμε, οτιδήποτε θεωρείς χρήσιμο, αλλά προς το πρώτο δεν μας έχεις δώσει τίποτα. Ελπίζω να απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι. Ευχαριστούμε κύριε Μασάντ. Κύριε Μασάντ, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων και προσβλέπουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα των ε, συζητήσεών σας με τον Επίτροπο κύριο Χίλ και όπως είδατε υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τη δική μας ε, πλευρά και εμείς έχουμε δώσει εντολή στην Κομισιόν εντολή να εξασφαλίσει ότι οι ανησυχίες σε ό,τι αφορά στο θέμα της ε, χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που προκύπτει από τη δράση μεγάλων χρηματοπιστωτικών παραγόνων πρέπει να αντιμετωπιστεί σωστά. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για την παρουσία σας και ελπίζουμε να τα ξαναπούμε σύντομα. Okay, thank you, colleagues. Now... Σας ευχαριστώ, συνάδελφοι. Πάμε στο επόμενο σημείο της συνέντησης διάταξης, ψηφοφορίες. Η έκθεση για την φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή ως προβλήματα για την, ε, για την προστασία σε αναπτυσσόμενες χώρες. Συμβασική τροπολογία Α. Ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές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 Δεν δουλεύει το μηχάνημα σας. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 22 με 26 απορρίπτεται. Τροπολογία 23. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. Συμβαστική C σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε έλεγχο για το δεύτερο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι την ίδια πλειοψηφία εγκρίνεται κανονικά, αλλά ας κάνουμε ένα έλεγχο, γιατί δεν βλέπω τα χέρια σας καλά. Άρχεται την ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική D. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 40 υπέρ κατά από... Νομίζω ότι απορρίπτεται. Ας κάνουμε έλεγχο για τροπολογία 40. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστή ή αγγλικό, ε, λατινικό υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται. Τροπολογία 42 υπέρ κατά αποχές απορρίζεται 43 υπέρ κατά αποχές απορρίζεται F συμβαστική σε τρία τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά νομίζω ότι εγκρίνεται θέλετε έλεγχο έλεγχος για το δεύτερο τμήμα Πέρας. Εγκρίνεται πράγματι. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Η ίδια πλειοψηφία εγκρίνεται. Συμβαστική G υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική I υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 63 υπέρ κατά έλεγχος. Για την τροπολογία 63 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική K υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική M υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική N σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Αλλά ας κάνουμε έλεγχο για το δεύτερο τμήμα. Συμβαστική N, Άρχιε την ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά <clears throat> αποχές εγκρίνεται. Με την ίδια συμβαστική O υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική P υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 97 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά Έλεγχο για το τμήμα τη 97. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται πράγματι. Το σύνολο του κειμένου όπως, όπως ε, έχει ε, ε, διατροποποιηθεί υπέρ κατά απόχες η έκθεση έχει εγκριθεί. Ναι, πρέπει να το κάνουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. 43 ψηφοί υπέρ, 2 κατά, 5 αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Πάμε στο επόμενο σημείο του Αντιπρόεδρου Πίτερ Σίμον. Ε, Πίτα Σίμον παίρνει την Προεδρία. χωρίς μικρόφωνο. <laughs> Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, σημείο 6. Έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για το σχέδιο γνωμοδότησης του κυρίου Κίρτσου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, Στρατηγικών Επενδύσεων και την διακυβέρνησή του. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στον εισηγητή πρώτα, ο κύριο Κίρσο. Σα Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω συντάξει αυτή τη γνωμοδότηση για την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων προ την Επιτροπή Περιφερειακών Θεμάτων για το Ταμείο ε, Επενδύσεων και την Οικονομική Διακυβέρνηση βάσει του άρθρου 23 του κοινού, του κοινού κανονισμού. Έχω ήδη λάβει σχόλια από τον συνάδελφό μας τον κύριο Φερνάντες Αλβάρες και επίσης αναμένω σχόλια από τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους συναδέλφους. Η υποθεσμία των τροπολογιών είναι 19 Μαΐου. Στη συνέχεια και εγώ μαζί με τους και οδησυσυγητές θα συναντηθούμε και για να καταλήξουμε σε ένα τελικό κείμενο για το σχέδιο γνωμοδότησης που να καλύπτει μόνο μία σελίδα ώστε να στείλουμε τα κατάλληλα πολιτικά μηνύματα. Το γενικό πλαίσιο της γνωμοδότησης είναι η αναγνώριση από εμά της σημασίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Διαρθρωτικών Επενδύσεων για να δώσει τις απαραίτητες επενδύσεις για την ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόλησεως το επενδυτικό περιβάλλον στην Ευρωζώνη σιγά σιγά βελτιώνεται και στη σύνολη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η σημασία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Διαθωτικών Επενδύσεων παραμένει. Θέλουμε επίση να ενισχύσουμε τη σύνδεση μεταξύ αυτού του Ταμείου με το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αν έχει κανείς το σωστό πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης, αν υπάρχει έλεγχος του προϋπολογισμού και του χρέους, τότε οι επενδύσεις είναι ευκολότερο να προσελκυστούν. Φυσικά υπάρχουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι εφαρμόζονται από την Κομισιόν και θα θέλαμε να εξασφαλίσουμε την εφαρμογή αυτών των κανόνων με την έννοια ότι αποδεχτόμεθα τη σχέση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Διαφορετικού και Επενδυτικού Ταμείου και του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης θα θέλαμε όμως να αποτρέψουμε να υπάρξουν προβλήματα, παραγωγός με τις ε, περιφέρειες ή κάποια επενδυτικά σχέδια να τύχουν να ουσιαστικά να τύχουν κυρώσεων, να, να χάσουν ε, τη δυνατότητά τους επειδή τα κεντρικά κράτη δεν έχουν ελέγξει το συνολικό τους έλλειμμα. Για το θέμα λοιπόν του επαναπρογραμματισμού αυτών των σχεδίων δεν θέλουμε να υπάρξει μια τέτοια διαδικασία, θέλουμε να την αποφύγουμε εάν είναι δυνατόν, και επίση να αποφύγουμε και την αναστολή πληρωμών. ενδεχομένω μπορεί να υπάρχουν κάποιε ακραίε καταστάσει οι οποίε μπορούν να οδηγήσουν σε τέτοιου είδου λήψη αποφάσεων. Εμεί θέλουμε, εν πάση περιπτώσει, να εμπλέξουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε θεσμικό επίπεδο στη διαδικασία λήψη αποφάσεων και θέλουμε επίση να δημιουργήσουμε και ένα σύστημα έγκαιρη προειδοποίηση αν ανακύψει κάποιο πρόβλημα για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά γιατί υποστηρίζουμε τις επενδύσεις και θέλουμε την ανάπτυξη των ε, περιφερειών και την οικονομική και κοινωνική συνοχή που είναι δύσκολοι στόχοι να επιτευχθούν. Αυτό είναι λοιπόν το κύριο κύρια κατεύθυνση της νομοδότησης. Ενδεχομένως ο κύριος Φερνάνδες Αλβάρης θα ήθελε να προσθέσει τα σχόλιά του. Είμαστε έτοιμοι για να ακούσουμε προτάσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κίλτσο δίνω καταρχήν το λόγο στον κύριο Φερνάντε Αλβάρε, ω κοιόδη για του σοσιαλιστέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχά θα ήθελα να αναγνωρίσω την προσπάθεια την οποία έκανε ο κύριος εισηγητής στα πλαίσια μιας γνωμοδότησης σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 23. Θα ήθελα να πω ότι το συγκεκριμένο άρθρο είχε καταψηφιστεί κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περίοδου από τη συγκεκριμένη Επιτροπή. Και γι' αυτό πέραν αυτού ε, εμείς ε, δεν μπορούμε παρά να σεβαστούμε τη νομική ρύθμιση. Το έγγραφο, εν πάση περιπτώσει, προσπαθεί να εξισορροπήσει κάπως την κατάσταση και είναι καλή ευκαιρία για να προχωρήσουμε στη συζήτηση των τροπολογιών τις επόμενες εβδομάδες. Θα ήθελα να κάνω τώρα δύο παρατηρήσεις, οι οποίες νομίζω είναι πολύ κοντά σε αυτά τα οποία λέει ο ίδιος ο εισηγητής. Η μακροαιρεσιμότητα και η πιθανή διακοπή της πρότασης η οποία ίσχυε είναι μια τελική αν θέλετε λύση, είναι μια λύση τελικής, η τελική ευκαιρία η οποία μπορεί να υπάρχει και θα πρέπει να ληφθεί εφόσον ληφθούν υπόψη μόνο οι συνέπειες οι κοινωνικές και οι οικονομικές. Η πάυση αυτή των πληρωμών, όπως είπαμε, είναι μια τελευταία επιλογή. Δεν θα πρέπει να χάσουμε ακριβώς την προοπτική που έχουμε του Ευρωπαίου πολίτη. Ο Ευρωπαίος πολίτης είναι το τελικό πρόσωπο το οποίο θα ωφεληθεί από την συγκεκριμένη αυτή ρύθμιση και θα πρέπει οι αποφάσεις οικονομικές να λαμβάνονται με σωστό τρόπο υπέρ του πολίτη. Και τώρα για τους Ευρωπαίους πολίτες οι οποίοι δεν έχουν την, την υπηκότητα της χώρας στην οποία κατοικούν θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα, δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις ε, εκλογές και χάνουν έτσι την ευκαιρία να ασκήσουν μια κάποια δυνατότητα πίεσης. Θα πρέπει λοιπόν τα διαφορετικά ταμεία να μας οδηγήσουν στο ε, να υπάρξουν οι κατάλληλες μορφές ε, επενδύσεων και να χρησιμοποιούνται τα κοινοτικά χρήματα σωστά. Ε, και να μην υπάρχουν καταχρήσεις. Το άρθρο 23 έμπαση περιπτώσει θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και είναι τελευταία λύση, αποτάτη λύση η διακοπή των πληρωμών. Θα πρέπει λοιπόν η, θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ενισχυθεί επίσης σε όλες τις φάσεις επεξεργασίας, προετοιμασίας, σύνταξης και στο τέλος να υπάρχει δυνατότητα έκφρασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στα πλαίσια που ε, ξεκινάει η διαδικασία που θα μπορούσε να καταλήξει σε απόφαση διακοπής των πληρωμών. Θα ήθελα λοιπόν στο τελικό κείμενο να υπογραμμίσουμε για μια ακόμη φορά ότι η πάυση των πληρωμών είναι μια τελική, μια απότατη λύση και θα πρέπει να υπάρξει μια πιο πρωταγωνιστική θέση ε, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Άλβαρες γιατί το ίσια ο Στανισλάβ Ούζοκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή που ετοίμασε ένα καλό σχέδιο κειμένου. Υποστηρίζω τις απόψεις του εισηγητή. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να τονίσω ότι το αίτημα για αναπρογραμματισμό των ταμείων με συνοδεία πολύ αυστηρών προϋποθέσεων δεν νομίζω ότι δημιουργεί πρόβλημα. Δεν δημιουργεί πρόβλημα και η προσφυγή στο άρθρο 23. Το βασικό όμω είναι να λάβουμε υπόψη την συνολική κατάσταση της χώρας και, της, ε, και των περιφερειών της. Με βάση την εμπειρία μας ξέρουμε ότι συχνά οι τοπικές αρχές θεωρούνται υπεύθυνε για τις δράσει της κεντρικής κυβέρνησης της χώρας. Επομένως, ζητάω από την ε, Κομισιόν να έχει μια πιο μακρόπνοη θεώρηση ε, σε περίπτωση που θέλει να προβεί σε αναστολή των πληρωμών ή σε περίπτωση που θέλει να αποσύρει κονδύλια. Από πλευρά μου τώρα θα ήθελα κάτι προσωπικό να πω. Χρειαζόμαστε διάλογο, χρειαζόμαστε διαφάνεια στην όλη διαδικασία. Αυτό είναι ένα προσωπικό σχόλιο. Ως, όπως είπε και ο ομιλητής, θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία. Και για να συνοψίσω, πιστεύω ότι χρειαζόμαστε περισσότερες διαφορετικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη-μέλη. Αυτό είναι μόνιμη από ομιλίας μου, το λέω πάντα. Μερσή, ε, κόρα για το, τους φιλελεύθερους. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το σχέδιο αυτογνωμοδότησης. Συμφωνώ με πολλά που λέει το σχέδιο γνωμοδότησης, ιδίω την ανάγκη να μειωθεί ο πολιτικός κίνδυνος για τους επενδυτές με την εξασφάλιση της σταθερότητας και προσβλέπω σε συνεργασία μαζί του και τους άλλους σκιώδεις συζητητές. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια και τι ευθύνε των κρατών μελών να μπορέσουν με σόφρονα τρόπο να δαπανίσουν τα χρήματα αυτά με τον τρόπο ο οποίος ενισχύει τη γενική του οικονομική δομή. Η Επιτροπή μας έχει τονίσει την σημασία της ενίσχυση τη ανταγωνιστικότητα και των αντιστοίχων δομών των κρατών μελών. Έχουμε τονίσει ότι οι περισσότερες συστάσεις ποτέ δεν εφαρμόζονται. Ούτε εν μέρη. Είδαμε τα τελευταία χρόνια ότι ορισμένα κράτη-μέλη έχουν παραγνωρίσει τις διάφορες συστάσεις για την οικονομική βελτίωση και τις συστάσεις αναχώρα. Το άρθρο 23 ως έχει δεν ενθαρρύνουν καθόλου τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσει και ανταμείβει τι χώρε, οι οποίε παρακάμπτουν τα διαρθρωτικά μέτρα. Βάσει του άρθρου 23, η Κομισιόν στην απόφαση τη αναστολή πληρωμών μπορεί να λάβει υπόψη μονάχα την οικονομική και κοινωνική κατάσταση στα κράτη-μέλη. Το άρθρο 23 συνδέεται επίση και με το παράδειγμα 3 που αναφέρει τα ποσοστά περικοπής τα οποία εξαρτώνται μονάχα από το ποσοστό ανεργία του αντίστοιχου κράτου. Αυτό δημιουργεί μια κατάσταση όπου τα κράτη-μέλη που έχουν αποτύχει να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσει και συστάσει. και επομένω έχουν υψηλό ποσοστό ανεργία, έχουν μικρότερα ποσοστά περικοπών. Ενώ τα κράτη-μέλη που έχουν ενισχύσει την οικονομία του και έχουν χαμηλότερη ανεργία βρίσκονται στην αντίθετη κατεύθυνση. Αυτό λοιπόν επιβραβεύει την μη συμμόρφωση και τιμωρεί την συμμόρφωση. Αυτό είναι ακατανόητο. Για να διορθωθεί αυτή η κατάσταση, η Κομισιόν όταν παίρνει αποφάσει για το πώ θα πρέπει να υπάρχουν αναστολέ πληρωμών, θα πρέπει να λάβει υπόψη και το ιστορικό κάθε χώρα στην εφαρμογή των καταχώρα χώρα ειδικών συστάσεων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχουν σωστά κίνητρα μείωση του ηθικού κινδύνου και ισοδίκαια μεταχείριση των κρατών μελών. Και πάλι κύριε Πρόεδρε, πώ βλέπω, στο να συνεργαστώ με τον εισηγητή ώστε να καταλήξουμε σε ένα αποτελεσματικό κείμενο ταχεία. Σας ευχαριστώ. Για την ΚΟΕ, ο κύριος Παπαδημούλης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εργασία που έχει κάνει μέχρι τώρα και θα ήθελα να θυμίσω σε όλους τους συναδέλφους όλων των πολιτικών ομάδων τη θέση που πήρε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέναντι στο άρθρο 23 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε μια θέση αρνητική, όπως σημείωσε και ο συνάδελφο από τους σοσιαλιστές. Εκτιμώντας ότι το άρθρο 23 υποβαθμίζει, υποβιβάζει τις πολιτικές συνοχής που είναι στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί θέτει περιορισμούς που οδηγούν στη διεύρυνση των ανισοτήτων και των κοινωνικών και των περιφερειακών θα υπερασπίσουμε αυτή τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ή θα πάμε business as usual από τη στιγμή που η Κομισιόν απέρριψε τη θέση του Ευρωκοινοβουλίου συμμορφωνόμαστε. Η θέση της πολιτικής μου ομάδας είναι ότι πρέπει να υπερασπίσουμε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να διεκδικήσουμε την ενεργοποίηση της παραγράφου 17 του άρθρου 23 που προβλέπει την επανεξέταση αυτού του άρθρου το οποίο ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί. Αλλά εκτός αυτού θα πρέπει να δούμε με βάση την κοινή λογική όχι πως θα αποδυναμωθούν κάποιες ρήτρε που έβαλε η Κομισιόν στην τελική πρόταση, όπως προτάθηκε από την προηγούμενη συνάδελφου, αλλά πως θα ενισχυθούν. Και αυτό περιμένω από τον εισηγητή να κάνει στην διαδικασία της διαβούλευσης με τους σκιώδεις εισηγητές. Να ενισχύσουμε το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως υπόθηκε. Να προστατεύσουμε τις περιφέρειες που δεν πρέπει να πληρώνουν την δημοσιονομική ασωτεία κυβερνήσεων να ενισχύσουμε προγράμματα που να στηρίζουν τη μείωση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων. Η πέμπτη έκθεση της συνοχής δείχνει ότι στα τελευταία χρόνια της κρίσης αυξήθηκαν και η ανεργία και η φτώχεια και οι περιφερειακές και οι κοινωνικές ανισότητες, μειώθηκαν οι επενδύσεις σε όλη την Ευρωζώνη και μειώθηκαν οι επενδύσεις στις χώρες που υποφέρουν από μεγαλύτερη ύφεση και μεγαλύτερη ανεργία. Δεν πρέπει η πολιτική συνοχής, η περιφερειακή πολιτική να ενισχύει αυτές τις ανισότητες. Θα πρότεινα στον εισηγητή να ε, αξιοποιήσει περισσότερο την έκθεση του κυρίου Λόπες που είναι ο βασικός εισηγητής εκ μέρους της Ρέτζη στην διαμόρφωση του τελικού σχεδίου γνωμοδότησης έτσι ώστε και να ενισχύσουμε παραπάνω το ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου στην όλη διαδικασία αλλά και να υπερασπίσουμε τις θέσεις που το Ευρωκοινοβούλιο υποστήριξε στη διάρκεια της προηγούμενης θητείας. Είμαι έτοιμος και με σχόλια και με τροπολογίες στην ε, περίοδο που θα ακολουθήσει να συμβάλλω σε αυτή την προσπάθεια αναζητώντας συνενέσεις προς αυτή την κατεύθυνση εφόσον και ο εισηγητής δείχνει ότι επιθυμεί να εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Δημήτρη. Ο Σβέν Γκίκολ για του πράσινου έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ για την έκθεση. Για το σχέδιο έκθεση συνάδελφοι. Εμείς ε, στην πατρίδα μου έχουμε διάφορα προβλήματα με τα μυρμήγκια. Το καλοκαίρι προσπαθούν να μπουν στο σπίτι σου και να φτιάξουν φωλιές. Το ξέρετε εσείς το πρόβλημα. Εάν θες να τα ξεφορτωθείς, έχει διάφορες επιλογές. Η μία επιλογή είναι να διαλύσει το σπίτι για να ξεπαστρέψει τις μυρμικοφολιές. Αυτό είναι λιγάκι το μέτρο που θέλουμε να λάβουμε εδώ. Και δεν το υποστηρίξαμε ούτε στην αρχή, γιατί το να αποσύρεις κονδύλια από περιοχές, ε, επιχειρήσεις και χώρες που έχουν ούτως ή άλλως προβλήματα, είναι σαν να θέλεις να δημιουργήσεις κίνητρα για να κάνεις καλή δημόσια πολιτική, αλλά στην πραγματικότητα ε, κάνεις μεγάλο κακό. Επομένως, συμφωνώ με τους συναδέλφους που ήταν επικριτικοί ως προς αυτή την προσέγγιση και επίσης είμαι απογοητευμένος που πολλοί ε, που πολλά κράτη-μέλη δεν ακολουθούν τις ειδικέ συστάσεις χώρα. Το ερώτημα είναι λοιπόν, είναι αυτό το σωστό όπλο για να καταπολεμήσουμε το πρόβλημα που έχουμε σε όλες τις χώρες, έτσι την, αν όχι σε όλες, σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενίσχυση λοιπόν της ε, γνωμοδότησης προς αυτή την κατεύθυνση είναι σημαντικό. Και να περιορίσουμε τη ζημιά που γίνεται λόγω αυτού. Το να προτείνουμε ένα καταλληλότερο όπλο για να υλοποιήσουμε το στόχο μας, καλό θα ήταν, έτσι, νομίζω. Τώρα, επί των λεπτομεριών. Υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο θα ήθελα να σκεφτούμε, παρότι συμφωνούμε με τη γενική προσέγγιση που υπάρχει στο σχέδιο έκθεσης. Για τους ειδικού τρόπους, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία που θα μας οδηγήσει στην αξιολόγηση που προβλέπεται στον κανονισμό των κοινών διατάξεων για τις, τη μακροαιρεσιμότητα που συνδέεται με, τα, με το Ταμείο Συνοχής. Το, η νομοθεσία που είχε υιοθετηθεί την προηγούμενη περίοδο προβλέπει μια τέτοια αξιολόγηση χωρίς όμως να μπαίνει σε λεπτομέρειες περαιτέρω ό,τι αφορά τη διαδικασία που θα μας βοηθήσει, χωρίς να μας ε, εξηγεί και την εμπλοκή ας πούμε, των stakeholders, των ενδιαφερομένων. Καλό θα ήταν, χρήσιμο θα ήταν να ρωτήσουμε την Κομισιόν να μας διευκρινίσει την αλληλεπίδραση ε, ανάμεσα στην πρόσφατη ε, ανακοίνωση για την ευελιξία και την ρήτρα με τις κατευθυντήριες γραμμές ε, μετά την ε, εκπόνηση του άρθρου 23 του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων. Οι πρόσωποι της Κομισιόν θα μπορούσαν ίσως να μας σχολιάσουν λιγάκι αυτό το... τη σχέση που υπάρχει, την αλληλεπίδραση ανάμεσα στις δύο διατάξεις. Ευχαριστώ Σβέν. Δεν ακοβάλει αυτό η ευθυντή. Ευχαριστώ. Συμφωνώ. Συμφωνώ με τους άλλους σκιώδεις εισηγητές ε, που ήταν επικριτικές προς αυτό το άρθρο 23, το οποίο θεωρούμε ότι και στην Επιτροπή Ρέτζη, ε, όπως υπόθηκε, πρέπει πολλά να αλλάξουν. Καταρχάς, το θέμα της ε, προσκόλλησης στους ε, κανόνες διακυβέρνησης. Αυτή είναι μια αρχή λανθασμένη εξυπαρχής. Ένα κράτος το οποίο δεν μπορεί να ε, σεβαστεί τους ε, κανόνες για τα ελλείμματα και το χρέος, έχει ανάγκη ακόμα μεγαλύτερη έχει ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη από τις πληρωμές. Το να σταματήσουμε, το να στείλουμε τις πληρωμές κατά 100% θα επιδεινώσουν τις ε, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Φυσικά σε περίπτωση απάτης ε, ή σε περίπτωση οργανωμένου εγκλήματος για τη χρήση των ταμείων, ναι, πρέπει να υπάρξει αναστολή. Πρέπει να πούμε ότι Έχουμε την αύξηση του ελλείμματος ε, σε εθνικό επίπεδο. Όμως, ε, αν εφαρμόσουμε το άρθρο 23, θα πληγούν οι περιφέρειες. Αυτό είναι παράδοξο. Επίσης, το αίτημα ε, αναπρογραμματισμού των συμβολέων επισύρει σημαντικό διοικητικό άχθος και αυτό θα το επομιστούν πάλι οι τοπικοί φορείς και οι περιφέρειες. Μία πρόταση που θα μπορούσαμε να κάνουμε για μεγαλύτερη ευελιξία είναι να αναθεωρήσουμε τη ρήτρα των επενδύσεων και τι θα γίνει με την, με την περιφερειακή συγχρηματοδότηση ή την εθνική συγχρηματοδότηση για να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να έχουν καλύτερη ε, ευελιξία. Είναι κάποιες προτάσεις που θα κάνουμε και ελπίζω να υπάρχει και δυνατότητα να βρούμε μια συμφωνία συμβιβαστική δεδομένου του ότι υπάρχει μια αρκετά πλατιά πλειοψηφία για να τροποποιήσουμε το άρθρο 23 προς την κατεύθυνση που λέμε. Μάρκο Βάλι. Ευχαριστώ τον Μάρκο Βάλι. Και τώρα υπάρχει ένας ε, που θέλει να λάβει το λόγο επιπλέον η κυρία Ήβα Μίλα. Μάλετη, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μας τον κύριο Γιώργο Κί, Κίρτσο για την έκθεση αυτή και χαίρομαι που ακούω ότι έχουμε κοινό στόχο όλοι, το να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μια συνεκτική εφαρμογή της πολιτικής συνοχής και να μην θέσουμε σε κίνδυνο τις αναπτυσσόμενες περιοχές μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά επιμένουμε για την καλή οικονομική διακυβέρνηση συγχρόνως και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και αυτά τα στοιχεία. Η καλή οικονομική διακυβέρνηση είναι μια προϋπόθεση για μια αποτελεσματική πολιτική συνοχής. Και Στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον υφιστάμενο κανονισμό. Νομίζω με τον τρόπο αυτό μπορούμε να δώσουμε καλά κίνητρα στα κράτη-μέλη να μην δουν την πολιτική συνοχή χωριστά από τις συνολικές τους οικονομικές πολιτικές που είναι μια συνήθις πρακτική αυτή τη στιγμή και μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει η πολιτική συνοχής να προχωρήσει από την απλή πολιτική επενδύσεω σε μια πολιτική ανάπτυξη. Χρειάζεται η πολιτική συνοχή να ατενιστεί ω πολιτική ανάπτυξη και όχι πολιτική επενδύσεων και μόνο. Συμφωνώ λοιπόν απόλυτα με την κυρία Κόρα ότι πρέπει να δούμε και την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής <clears throat> των ειδικών αναχώρα συστάσεων και ότι οι μακροοικονομικοί δείκτες θα μπορούσαν ίσως να τροποποιηθούν και η Κομισιόν θα πρέπει να λάβει περισσότερο η υπόψη της τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες μέλη έχουν εφαρμόσει τις ειδικές αναχώρα συστάσεις και σε επίπεδο σχεδιασμού και στα λειτουργικά σχέδιά τους και στις εταιρικέ σχέσεις και επίσης να αναλύσουν και την εφαρμογή των λειτουργικών προγραμμάτων στην πράξη και κατά πόσο όλα αυτά συνάδουν με τις ειδικές αναχώρα συστάσεις. Χαίρομαι που μπορώ να συμμεριστώ μαζί σας. Πληροφορίες που έλαβα από την Κομισιόν μου είπαν <clears throat> ότι τώρα έχουν μπει στη διαδικασία ανάλυσης του κατά πόσον τα κράτη-μέλη έχουν λάβει υπόψη τους στα λειτουργικά τους προγράμματα τις ειδικέ αναχώρα συστάσεις. Έτσι, η Κομισιόν θα προετοιμάσει ένα έγγραφο στο οποίο θα απεικονίζεται και θα αναλύεται η συμμόρφωση προς τις ειδικέ αναχώρα <clears throat> συστάσεις με τις ε, προτεραιότητες και τις δράσεις των λειτουργικών προγραμμάτων και θα παρακολουθήσουν στη συνέχεια και την εφαρμογή όλων αυτών των ενέργειών που θα πρέπει να εντάσσονται στα λειτουργικά προγράμματα και με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η απαραίτητη σύνδεση μεταξύ της ε, πολιτικής συνοχής και της οικονομικής ευκυβερνησίας. Θα ήθελα όμως επιπλέον να καταγράψω και ένα σημαντικό πρόγραμμα που και αυτό συνάπτεται με την οικονομική ευκυβερνησία. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει συζητηθεί πολλές φορές στην Επιτροπή Προϋπολογισμού και την Περιφερειακή Επιτροπή, αλλά δεν έχει ανακύψει στη δική μας Επιτροπή παρά τη σημασία που έχει. Είναι τα μη εκταμιευθέντα ποσά από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Έχουμε καθυστερήσει τα μάλα για την εκταμείευση ποσών για την πολιτική συνοχή, αλλά όχι μονάχα και για άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό σημαίνει ότι έχουμε πρόβλημα με την σωστή οικονομική διακυβέρνηση. Γιατί υπάρχει και μια οδηγία που εφαρμόζει χρονικά όρια για την καταβολή των ποσών. Λέει ότι μέχρι, ε, σε, μέχρι το όριο των 60 ημερών θα πρέπει να καταβληθούν όλε τι υποχρεώσει από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο δεν πράττει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Είναι απαραίτητο λοιπόν ότι δεν θα είναι μονάχα αυτέ οι δύο επιτροπέ που άπτονται του θέματο αυτού, αλλά και εμεί ω η Επιτροπή Αρμόδια για την Καλή Οικονομική Διακυβέρνηση να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ιβάνα. Βλέπω, μη βλέπων άλλον ο οποίο θέλει να λάβει το λόγο προς το παρόν και επομένως θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Κομισιόν εφόσον θέλει να παρουσιάσει τη δική της άποψη. Ja, das ist der Fall. Bitte ε, Thank you very much, Mr. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχω να κάνω πολλές παρατηρήσεις από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την δουλειά την οποία έχει προετοιμάσει η σύνδεση ανάμεσα στη χρηματοδότηση την κοινοτική από τη μία και την χρηστή οικονομική διακυβέρνηση από την άλλη, η σύνδεση αυτή είναι καθοριστική. Και γι' αυτό ακριβώς έχουμε εμείνει σε συγκεκριμένες προτάσεις στα πλαίσια του νέου νομικού πλαισίου. Θεωρώ ότι η αποτελεσματικότητα της κοινοτικής επένδυσης ισχύει μόνο στα πλαίσια ενός μακροοικονομικού περιβάλλοντος υγιούς ε, ίσως κάποιες μικρές διευκρινήσεις. Καταρχάς θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, <clears throat> θα μπορεί να διαβουλεύεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, σε όλες τις περιπτώσεις της εφαρμογής αυτών των ρυθμίσεων για την μακροαιρεσιμότητα. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώνουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πιθανές διακοπές πληρωμών και για μη αποτελεσματικές δράσεις και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα είτε την εκκίνηση ενός διαρθρωμένου διαλόγου είτε την απλή λήψη υπόψη των, της γνώμης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πάνω σε θέματα τα οποία εμείς θα προτείνουμε. Η σύνδεση επίσης ανάμεσα στις ρυθμίσεις για την μακροοικονομική αρεσιμότητα και από την άλλη αυτή η συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει για την ευελιξία ε, του Συμφώνου Σταθερότητας. Θα ήθελα να τα διευκρινίσω αυτά τα δύο λιγάκι. Γιατί στα πλαίσια της μακροαιρεσιμότητας και των ρυθμίσεων της μακροαιρεσιμότητας οι κανόνες είναι σαφείς. Εφόσον μια χώρα μπει σε μια διαδικασία υπερβολικού χρέους, σε μια διαδικασία δηλαδή μακροοικονομικής έλλειψης σταθερότητας και εφόσον δεν ακολουθεί τις συστάσεις τις οποίες λαμβάνει από το Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να διακόψει την χρηματοδότηση. Υπάρχει σχεδόν ένας κάποιος αυτοματισμός εδώ. Μιλάμε για χώρες οι οποίες είναι στα πλαίσια του λεγόμενου διαρθρωτικού τμήματος του Συμφώνου Σταθεροποίησης. Διορθωτικού, συγγνώμη, ε, τμήματος Είχαμε το Φεβάριο μιλήσει και για τα θέματα ευελιξίας και υπάρχει η λεγόμενη επενδυτική ρήτρα. Η επενδυτική ρήτρα αφορά την εθνική συγχρηματοδότηση των κοινοτικών προγραμμάτων. Μπορεί κανείς να τραβήξει τα, τις πιστώσεις αυτές εφόσον βέβαια έχει τη δυνατότητα να συγχρηματοδοτήσει σε εθνικό επίπεδο. Αυτό είναι, ένα, είναι κάτι το οποίο περιλαμβάνεται στο έλλειμμα ε, των χωρών. Τώρα, για τις χώρες που είναι στο προληπτικό τμήμα του συμφώνου, όχι στο διορθωτικό, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, οι χώρες αυτές μπορούν να ζητήσουν για μία προσωρινή εξέρεξη από τον, από τον κανόνα αυτό. Ότι δηλαδή η εθνική συγχρηματοδότηση για τα κοινοτικά προγράμματα θα αφαιρεθεί από το δημοσιονομικό έλλειμμα, αλλά μόνο σε προσωρινή βάση δίδει αν θέλετε κάποιο περιθώριο αναπνοής για συμπληρωματικές επενδύσεις. Αυτή ήταν μια διευκρίνηση. Κατά τα άλλα δεν έχω να πω κάτι. Σας ευχαριστώ για τις διευκρινήσεις αυτές. Τέλος, ο εισηγητής έχει και πάλι το λόγο για να κάνει μια σύνοψη. Ε, well, I would like to... Θέλω να ευχαριστήσω τους αδέλφους για τα ενδιαφέροντα σχόλιά τους και τις υποδείξεις τους. Νομίζω ότι είναι συγκλίνοντα τα σχόλια. Εγώ είμαι υπέρ μιας βαθμίας προσέγγισης προσωπικά. Θα δούμε όμως τι θα συμβεί, θα το συζητήσουμε. Θα ήθελα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βοηθήσει με τη συμμετοχή του στον έλεγχο της διαδικασίας να συμμετάσχει στη διαδικασία που περιγράφτηκε παρά να έχουμε ένα πόλεμο ας πούμε παραθέσεων και αντιπαραθέσεων ε, μεταξύ Κομισιών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περιμένω να γίνει λοιπόν μια επικοδομητική συζήτηση με τους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Η προθεσμία για τροπολογίες είναι η 19η 9 η Μαΐου στις 5 το απόγευμα η συζήτηση για τις τροφολογίες στις 16 Ιουνίου και θα ακολουθήσει και η ψηφοφορία στις 25 Ιουνίου. Η αρμόδια επιτροπή Ρέγγι θα ψηφίσει στις 13 και 14 Ιουλίου, τουλάχιστον με τον τωρινό σχεδιασμό. Σημείο 13, διάφορα θέματα. Υπάρχει κάποιο άλλο θέμα που θέλετε να γίνετε, εάν όχι Απλώς σας πεθυμίζω ότι η επόμενη συνεδρίασή μας θα γίνει την 3η 26 Μαΐου 15 με 18 και 30. Και τώρα μου λένε όχι, όχι, όχι. Παρακαλώ τη γραμματεία να μου πει γιατί όχι, όχι, όχι. Πότε είναι η επόμενη μας συνεδρίαση. Φυσικά. 26 Μαΐου αλλά σας υπενθυμίσω ότι αύριο έχουμε την ανταλλαγή απόψε με τον κύριο Μίσελ Σαπέν και παρακαλώ τους συναδέλφους να είναι παρόντες. Ευχαριστώ πολύ που μείνατε ως το τέλος και σας εύχομαι καλό απόγευμα.